you ready? Can, can, we, can we start? Um, welcome back to this afternoon session. a few minutes late. Να ξεκινήσουμε, ε, ε, γιατί έχουμε πολλά να καλύψουμε και έχουν περάσει λίγα λεπτά ήδη. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων για τις ε, τροπολογίες για τη, έκθεση, για τη διακυβέρνηση της ενέας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015. Η συγγήτρια είναι η κυρία Γκάλ Πέλτς. Συγγνώμη αν δεν προφέρω σωστά το όνομά σας. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τις τροπολογίες ε, και αν κάποιος ε, δεν είναι στον κατάλογο των σχεδόν εισηγητών και θέλει να μιλήσει, παρακαλώ να λάβετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδης εισηγητές καθώς και άλλους συναδέλφους για τη συνεργασία τους μέχρι τούδε. Η συνεργασία αυτή ήταν ε, ιδιαίτερα επιτυχής, δεδομένου ότι είχαμε και πολύ σύντομες προθεσμίες και παρά το γεγονός ότι μας πίεζε ο χρόνος, οι συνάδελφοι ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι και κατέθεσαν 161 τροπολογίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γεγονός που σημαίνει ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι συνάδελφοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα ε, για τα όσα κάνω. Οι περισσότερες από τις τροπολογίες συνάδουν με το αρχικό σκεπτικό μου και αυτό φυσικά με διευκόλυνε ιδιαίτερα. Υπάρχει σύμπτωση απόψεων και οι περισσότεροι συνάδελφοι συμφωνούν ή μάλλον όλοι συμφωνούν ότι προκειμένου να λειτουργεί καταλήλωση η νέα αγορά χρειαζόμαστε πρέπει να προσέξουμε καλύτερα την εφαρμογή ε, του νομικού πλαισίου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα και προσκόμματα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα και να άρουμε τα προσκόμματα. Όσον αφορά τα καθήκοντά μας, το ρόλο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Πρέπει να δούμε πού έχει επιτευχθεί πρόοδος και θα πρέπει επίσης να εντοπίσουμε τις δυσκολίες. Να σας παραπέμψω και σε κάτι δυσάρεστο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ετοιμάσει κάποιο έγγραφο για την ολοκλήρωση της ενίας αγοράς, τον οποίο, το οποίο να συνοδεύει την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης. Θεωρώ ότι είναι λυπηρό το γεγονός αυτό και θα ήθελα να μου πούν γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο φέτος και γιατί ακολουθούμε διαφορετική δομή. Θα ήθελα να μου το εξηγήσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί άλλαξε η προσέγγιση τους φέτος. Και θα ήθελα να υποβάλω και μία τροπολογία, ελπίζω να την υποστηρίξουν οι περισσότεροι συνάδελφοι, ε, για να διορθωθεί αυτό. Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες, με χαρά μου διαπιστώνω ότι οι περισσότερες τροπολογίες επικεντρώθηκαν σε ε, συγκεκριμένους τομείς ιδιαίτερη σημασία, στους οποίους υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης. Ε, δίκτυα, ψηφιακή οικονομία, οι τροπολογίες, όπως και η αρχική έκθεση, καταρχάς επισημαίνουν την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί και εκφράζουν και την επιθυμία να χρησιμοποιήσουμε το, τις δυνατότητες που μας προσφέρουν αυτές οι υπηρεσίες. Η ενιαία αγορά είναι πολύ καλή όσον αφορά τα αγαθά, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει και κατάλληλο ε, νομικό πλαίσιο για αυτό τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο και για τις υπηρεσίες. Καλωσορίζω τις τροπολογίες που θέλουν να βελτιώσουν τη λειτουργία του ε, οικονομικού τομέα, του χρηματοπιστωτικού τομέα και φυσικά τις υποστηρίζω αυτές τις τροπολογίες. Οι συνάδελφοι υπέβαλαν τροπολογίες και για την ψηφιακή έννοια αγορά. Μπορώ να υποστηρίξω τις περισσότερες τροπολογίες, διότι θεωρώ ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλήρως ε, τις δυνατότητες ε, που δεν έχουμε ακόμα χρησιμοποιήσει στον τομέα αυτό. Και τα δίκτυα εξακολουθούν να είναι εξίσου σημαντικά και είναι και η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην ε, ε, ανακοίνωση ε, e-communication για την ενέργεια και τις μεταφορές. είναι 8,5% προστιθέμενης αξίας και καλύπτουν το 6,1% της απασχόλησης οι τομείς αυτοί. Ο ψηφιακός τομέας αποτελεί κινητήριο μοχλό της παραγωγικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Οι τροπολογίες για το συγκεκριμένο ζήτημα, την ψηφιακή οικονομία, υποστηρίζονται από πλευρά μου. Μπορεί να χρειαστεί βέβαια να γίνουν και κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες γιατί υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις. Θα ήθελα να ε, σταθώ σε κάποιες τροπολογίες τώρα. Να ξεκινήσω με την ε, τροπολογία 15 των κυρίων Κοφεράτη και Γκουτιέρεθ, οι οποίοι ζητούν να υπάρξει μια πολιτική επανακβιομηχάνησης, μια στρατηγική ε, σε για κομβικούς τομείς ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μας. Η άποψή μου είναι ότι η τροπολογία αυτή σε κάποιο βαθμό είναι εκτός πεδίου εφαρμογής ε, της έκθεσής μου. Είναι αμφισβητήσιμο το κατά πόσον υπάρχει προστιθέμενη αξία, κυρίως για την ενή αγορά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να την ξαναδούμε με τους συναδέλφους και να το συζητήσουμε το ζήτημα αυτό. Ε, η πρώτη μου όμως αντίδραση είναι ότι η τροπολογία αυτή είναι εκτός ε, πεδίου εφαρμογής της έκθεσής μου. Ε, μια άλλη τροπολογία στην οποία θα ήθελα να σταθώ είναι μια τροπολογία η οποία καλύπτει ένα πολύ σημαντικό τομέα και το συζητούσαμε και στο Στρασβούργο. Την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της, φορο... και της απάτης, της φορολογικής απάτης. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό μεν, αλλά ο τρόπος με τον οποίο είναι διατυπωμένη δεν είναι ο κατάλληλος, διότι μπορεί να δημιουργήσει πεδίο για ε, συγκρούσεις και νέες πολιτικές συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται εδώ στην έκθεση αυτή ε, να καταγγέλουμε πολιτικούς ή χώρες. Όσον αφορά τη λειτουργία των μέτρων για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, και παρά το γεγονός ότι συμφωνώ με τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση, έχω κάποιες επιφυλάξεις ε, για κάποιες εξ αυτών. Ναι, Τις τροπολογίες 42 και 43 τώρα θα σας σχολιάσω. Το πρόβλημα μου είναι ότι θεωρώ ότι οι τροπολογίες αυτές είναι αμφίσιμες. ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει τη δυνατότητα να παρουσιάζονται οι συγκεκριμένες εκθέσεις αναχώρα πριν από την έγκρισή τους από το Συμβούλιο στα Εθνικά Κοινοβούλια. Θεωρώ ότι η ε, εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι λίγο αμφισβητήσιμη και κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει συζήτηση από του ζητήματος. Υπάρχει στη συνέχεια μια τροπολογία που ζητάει ε, εκθέσεις ανατρίμηνο. Ε, θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό, δεν ε, ε, είναι πρακτικό άλλωστε. Πρόκειται όμως για ένα από τα ζητήματα που θα ήθελα να συζητήσω με τους κοιόδης συζητητές. Κύριε Πρόεδρε, αυτά περιληπτικά για κάποιες από τις τροπολογίες που κατέθεσαν οι συνάδελφοι. Όπως σας είπα, στην πλειονότητά τους ε, συνάδουν με τη γενική μου προσέγγιση, με την εξαίρεση αυτών που σας επεσήμανα, όπου θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει κάποια περαιτέρω συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στη συνεχή μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Sergio Gutierrez. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εισηγήτρια, για την τοποθετήθε και για την εργασία που επιτέλεσε σε κλίμα κατανόησης και θετικό. Θα ήθελα αρχίζοντας να πω ότι θα πρέπει ως Επιτροπή ΙΜΚΟ να τοποθετηθούμε σε σχέση με κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι κάτι για το οποίο έχουμε καθυστερήσει. Στα πλαίσια της διαδικασία του πρώτου εξαμήνου δεν υπάρχει έκθεση για το θέμα που μας απασχολεί. Πρόκειται για ένα βήμα προς τα πίσω και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Το σύνολο της Επιτροπής μας και το Προεδρείο θα πρέπει να απευθυνθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή ώστε για το συγκεκριμένο θέμα να προτείνει μια διόρθωση για να μην ξανασυμβεί και πάλι. Κατανοώ ότι σε αυτό το νέο στάδιο που βρισκόμαστε να έχουμε την οικονομική ανάπτυξη και έχουμε βαρεθεί να ακούμε ότι η προτεραιότητα είναι η οικονομική ανάπτυξη και να βλέπουμε ότι δεν ακολουθούνται οι κατάλληλες πολιτικές αηφόρος ανάπτυξη, αλλά διαφορετική από ό,τι τα τελευταία χρόνια. Πλαίσια της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και της ψηφιακή αγοράς. Υπάρχει λοιπόν αντίθεση μεταξύ αυτών το οποίο λέγει η Κομισιόν και αυτά τα οποία αναφέρονται στη προσάρτημα όπου δεν γίνεται αναφορά στην οικονομική ανάπτυξη. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να το επισημάνει η Επιτροπή μας. Γιατί τελικά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι το μόνο μέσο και η μόνη διαδικασία που διαθέτουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα γενικότερα ώστε να μπορέσουμε στα πλαίσια του ε, Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως και τα κράτη-μέλη, να κάνουμε διορθωτικές Φράσεις, Διότι τώρα υπάρχει μια νέα οικονομική στρατηγική την οποία θέλει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει η Επιτροπή και να δούμε πώς με τις ειδικέ συστάσεις, ειδικέ συστάσεις σε ένα χώρα, με τις ε, αιτήσει εκθέσεις για οικονομική ανάπτυξη σε κάθε χώρα και σε σχέση με τις προηγούμενες προτάσεις τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Επίσης υπάρχει μια έλλειψη όθησης. Πολλές φορές λέγεται αυτό μια κόποση από τις διαφορετικές αναθεωρήσεις τις οποίες θέλουμε να κάνουμε στις πολιτικές μας. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε υπέρ της εσωτερικής ψηφιακής αγοράς, της οικονομικής ανάπτυξης γενικότερα, ώστε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και όχι περικοπές όλο και περισσότερους προπολογισμού. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει, όπως λέγω, όλα αυτά τα θέματα να τα λάβουμε πολύ σοβαρά στα πλαίσια της διαδικασίας του ευρωπαϊκού ε, εξαμήνου και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Επιτροπή να πούμε στην Επιτροπή ότι πρέπει να διορθώσει την γραμμή πλοήγησής της. Το σύνολο των ομάδων παρουσίασαν τροπολογίες οι οποίες είναι συνεκτικές. Τα φυσικά όντως θέλουμε να προχωρήσουμε προς την κρίση της εσωτερικής αγοράς, της πραγματικής. Υπάρχουν σε συγκεκριμένες τροπολογίες διαφορετικά σημεία, διαφορετικές προτεραιότητες όσον αφορά το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά σε γενικές γραμμές συμφωνούμε. Υπάρχει όμω μία τροπολογία που με απασχολεί που θέλει να αποτελέσει τροχοπέδι στην ενιοποίηση της ενία εσωτερικής αγοράς. Πρόκειται για τροπολογία με την οποία είμαστε εντελώ αντίθετοι. Πιστεύω όμω ότι κατά τα άλλα θα πρέπει να καταλήξουμε στις περισσότερε τροπολογίε με συνένεση ώστε να έχουμε μία πάρα πολύ ε, παγιωμένη και γενική θέση. Οι προτάσει μας σχέση με την πρόταση Επιτροπής, οι προτάσεις μας Νομίζω και οι προτεραιότητε μα διορίζονται σωστά. Αυτό που θέλουμε πρώτα απ' όλα είναι να επεφεληθούμε από τα σχέδια επενδύσεων όπω Φερρυπίν, το σχέδιο Juncker με τις ε, περιορισμούς του και με τα ε, προβλήματα που έχει. Νομίζω ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι επωφελείς σε διάφορους τομείς, κυρίως στον ενεργειακό τομέα, στον εξαρτώμεθα στα ενεργειακά λιγότερο από τρίτες χώρες να μειώσουμε στον τομέα αυτό το κόστος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Θα, θέλω, θα ήθελα επίσης να δούμε από κοντά περισσότερο διάφορα πάγιε, να δούμε διάφορες πάγιες δαπάνες κάποιων επιχειρήσεων. Ξέρουμε πολλές φορές ότι οι πάγιες δαπάνες προσωπικού δεν αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, ενώ οι ενεργειακές δαπάνες είναι κατά εκατοντάδες ποσοστά ε, ανώτερες τώρα τελευταία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια πραγματικά ενιαία ενεργειακή ευρωπαϊκή αγορά ώστε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να μειωθούν οι ενεργειακές δαπάνες των επιχειρήσεων μας. Επίσης θα ήθελα να κάνουμε επενδύσεις εξ από την ενεργεία στην ψηφιακή οικονομία και σε όλα τα έργα υποδομής που είναι απαραίτητα για να έχουμε μια πραγματικά ενιαία εσωτερική αγορά. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης πραγματικά να έχουμε ως έναν από τους κύριους στόχο μας στην ψηφιακή ενιαία εσωτερική αγορά. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση, δεν παίρνουμε τα πράγματα σοβαρά διαφορές μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τρομερά και νομίζω ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι εύκολα προσβάσιμο και όχι πολύ δαπανηρό και θα πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε να υποφεληθούν όλες οι επιχειρήσεις, οι μία και οι μεγαλύτερες, διότι αν δεν έχουμε μία ενιαία εσωτερική ψηφιακή αγορά, διότι δεν έχουμε τα καλά τα άλλα ενάβσματα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Επίσης, μιλάμε για επαναβιομηχανοποίηση, αυτός είναι ένας κοινό παρανομαστής και για την ανταγωνιστικότητα και δεν είναι αρνητικό για τον ανταγωνισμό. Έχουμε διαφορετικές ε, βιομηχανίες σε διάφορους τομείς και τώρα μιλούμε για την ψηφιακή ε, βιομηχανία και σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου η βαρύτητα του βιομηχανικού τομέα είναι μόνο της τάξης του 2,5%. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε καθυστέρηση πολλών ετών, αλλά θα πρέπει να κάνουμε σχέδια αναθεώρησης και ανάπακ, ε, ανάκαμψης. Δεν χρειάζεται πάντα στην ε, ε, να θέλουμε να γυρίζουμε πίσω στην σιδηροβιομηχανία. Υπάρχουν και άλλες αγορές που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, αλλά δεν υπάρχει κανένα στρατηγικό πρόγραμμα ή σχέδιο ή σχεδιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας το πάρουμε αυτό σοβαρά υπόψη. Υπάρχουν ε, στο σύνολο των ε, Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά προβλήματα στον τομέα αυτό και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Πιστεύω επίσης ότι την ε, διασυνοριακή ε, παραγωγή, τις κοινέ υπηρεσίες, τις ε, δημόσιες κοινοπραξίες, τους συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων στους πληστηριασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που θα προσδώσει συμπληρωματική αξία στην βιομηχανία μας. Το 99% των επιχειρήσεων συμμετέχουν μόνο σε μειοδοτικούς και δημόσιους διαγωνισμούς στη χώρα τους. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να επωφεληθούμε και από την ενιαία εσωτερική αγορά συμμετέχοντας και σε ε, μειοδοτικούς διαγωνισμούς άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν ότι αν έχουμε την δώσουμε την κατάλληλη όθηση θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ε, ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, να βοηθήσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας με θετικό τρόπο. Θα ήθελα να τελειώσω εδώ ευχαριστώντας και πάλι την ε, εισηγήτρια για την ε, εργασία που επιτέλεσε για την διάθεσή της να είναι σε συνεχή διάλογο και ελπίζω ότι ακόμη μια φορά θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτή την επιστοδρόμηση που διαπιστώνουμε στις προσθέσεις της Επιτροπής όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη στα πλαίσια της νέας εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. για την ECR Σκιώδης. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στο θέμα του εξαμήνου των στόχων και πώς θα παραμείνουμε ε, πιστοί σε έναν σημαντικό στόχο που είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και ότι δεν θα επιβληθεί κάτι από πάνω προς τα κάτω και ότι θα διατηρήσουμε ένα σχετικά ε, υψηλό ποσοστό ευελιξίας στη συνεργασία μας. Βεβαίως, οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μπορεί να είναι και άλλου είδους και για πολλούς τομείς δεν έχουμε δείκτες. Σε κάποιους έχουμε, σε κάποιους δεν έχουμε. Και θα πρέπει όλοι αυτοί οι δείκτες που διαθέτουμε να χρησιμοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, να επιλέξουμε δείκτες που ουσιαστικά μετρούν την ευρωπαϊκή αποδοτικότητα, τις ευρωπαϊκές επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη εικόνα της ευρωπαϊκής αγοράς και οικονομίας. Και βλέπω επίσης ότι έχουν υποβληθεί τροπολογίες και για την ε, ανταγωνιστικότητα συνολικά επίσης για τις λεπτομέρειες ε, της διαβούλευσης που έλαβε χώρα και της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων ε, σε αυτήν. Άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Πιστεύω πραγματικά ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία επιλογής της καλύτερης δυνατής ρύθμισης. Και εγώ θα υποβάλω τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ο τομέας της ενέργειας, σίγουρα εδώ θα πρέπει να επιτευχθούν δύσκολες περίπλοκες συμβαστικές λύσεις. Ο τομέας των υπηρεσιών, άλλη τροπολογία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, e-commerce. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα θέμα, όχι μόνο το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να παραμείνει σαν τομέας μέσα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι προστατεύοντας τον τομέα αυτό προστατεύουμε μόνο τις ελεύθερες συναλλαγές, το εμπόριο, αλλά και την τεχνολογία, την καινοτομία, τις νέες εφευρέσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να προστατεύσουμε τον τομέα αυτό με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική και σκληρή σας εργασία, αλλά πιστεύω ότι καλό θα ήταν σε πολλά από αυτά τα σημεία να βρούμε συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Η ομάδα των φιλελευθέρων. Καταρχήν, να επιστήσω την προσοχή σας στις τροπολογίες της δικής μας πολιτικής ομάδας των φιλελευθέρων. Το θέμα της μεθοδολογίας για την καταμέτρηση, τη μέτρηση των μειώσεων. Πώς το κάνουμε, υπάρχει μεθοδολογία, διότι πρέπει να μετρηθούν αυτές οι περικοπές. Βέβαια όλα αυτά είναι πολύ βαριές και επίπονες διαδικασίες για κάποιες ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάποια κράτη-μέλη κάτι έχουν κάνει, αλλά εδώ θα πρέπει να συγκρίνουμε τις εθνικές ε, πρακτικές και να επιλέξουμε την καλύτερη. Και γι' αυτό και εδώ θέτω το θέμα της μεθοδολογίας. Δεύτερον, η υλοποίηση του ευρωπαϊκού εξαμήνου ναι, πήραμε την απόφαση, τώρα πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή. Και προτείνω εδώ το ψήφισμα της 14ης Οκτωβρίου της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω ότι ε, και αυτό κάνω στην τροπολογία 43 θα υιοθετήσουμε όλη αυτή την διατύπωση. Η λειτουργία, η σωστή λειτουργία της ε, Ενίας αγοράς είναι κάτι το οποίο σαφώς και θα διευκολύνει τους επενδυτές. Τους επενδυτές και τους καταναλωτές, οι οποίοι πλήττονται σήμερα από τον κατακαιρματισμό αυτής της ενιαίας αγοράς. Και την ίδια ώρα χρειαζόμαστε και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να επανέλθει η εμπιστοσύνη, να περάσουμε από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να επανέλθει η εμπιστοσύνη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο τομέας της ψηφιακής ε, οικονομίας, εκεί όπου πάσχουμε σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείες και εδώ αναφέρομαι βεβαίως και σε άλλες τεχνολογικές ε, επιτυχίες όπως το χάρη το τα 4G τα οποία θα πρέπει να γενικευθούν παντού. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε πραγματικά μια ψηφιακή ενιαία αγορά στην Ευρώπη. Υπάρχουν τρόποι, πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, γιατί τα κείμενα μεν υπάρχουν, στην πράξη όμως δεν λειτουργεί το σύστημα και πρέπει να βελτιώσουμε εδώ την προστασία αυτή, προσδίδοντας ε, νέες το δυναμικό της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής οικονομίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι πολύ μεγάλο. Και την ίδια ώρα θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, η δημόσια δίκη της Ευρώπης θα γίνει πιο αποτελεσματική, πιο γρήγορη και πιο οικονομική. Ευχαριστώ πολύ δεν ιστιών. Ευχαριστώ πολύ Βίκη. Ευχαριστώ γιατί πραγματικά θεωρώ ότι το σχέδιο έκθεση αυτό είναι εξαιρετικό και συμφωνώ με όλους όσους πήραν το λόγο και μίλησαν για την ψηφιακή ενιαία αγορά δεν έχω υποβάλει πολλές τροπολογίες προς αυτή την κατάφτυνση, αλλά ακούγοντας όλα αυτά για τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν στο τομέα αυτό και για τα δικαιώματα των καταναλωτών με βρίσκουν σύμφωνο. Δεν θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε απλώς τους επενδυτές, αλλά χρειαζόμαστε και την ευρεία υποστήριξη των Ευρωπαίων πολιτών. Τα προβλήματα που σήμερα πλήττουν ε, τους Ευρωπαίους πολίτες πτώχεια, ανεργία, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, την εμπιστοσύνη προς την ευρωπαϊκή οικονομία και βλέπετε τις τάσεις που διαγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας αυτής της ανεργίας και των προβλημάτων στην αγορά. Θεωρώ λοιπόν ότι οτιδήποτε υπονομεύει εδώ τις αρχές της ενέας αγοράς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Οι τροπολογίες λοιπόν που ενισχύουν αυτές τις πτυχές είναι κατά την άποψή μου σωστές. Δεν υπάρχουν πολλά επαναστατικά στοιχεία και νέες ιδέες ε, σε αυτές τις προτάσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν είναι και η πρώτη φορά που μας απασχολεί. Το θέμα του TTIP τώρα, της ε, εμπορικής ε, συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θέλω τώρα εδώ να μπούμε στη γενική συζήτηση αν είναι κάτι καλό ή κακό. Πιστεύω όμως ότι όσον αφορά τη δική μας Επιτροπή είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το θέμα της συνεργασίας σε ρυθμιστικό επίπεδο. Δηλαδή, όταν πρόκειται για συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, θα πρέπει να ξαναδούμε τις παλιές αποφάσεις, τους παλιούς κανονισμούς και ρυθμίσεις και το Κοινοβούλιο δεν εκπροσωπείται στο Συμβούλιο για τα ρυθμιστικά θέματα. Θα υπάρξουν λοιπόν κάποιες διαπραγματεύσεις ως συνήθως μεταξύ κάποιων υψηλόβαθμων υπαλλήλων της Επιτροπής. Θα υπάρξουν συμφωνίες όπως αυτή που έχει υπογραφεί με τον Καναδά. Το αποτέλεσμα θα μας υποβληθεί και εμείς καλούμεθα στην τελική φάση να πούμε ναι ή όχι. Τι νόημα έχει να έχουμε εδώ στο Κοινοβούλιο μία αρμόδια επιτροπή για θέματα εσωτερικής αγοράς και να μην μπορούμε να παρέμβουμε σε ένα πιο έγκαιρο στάδιο. Ερωτώ λοιπόν την Επιτροπή πώς μπορούμε εδώ να υιοθετήσουμε μια διαφορετική διαδικασία καθότι το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών και το Κοινοβούλιο του Καναδά εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους. Εμείς όχι. Θα ξαναπάρω το λόγο γιατί θεωρώ ότι το θέμα της ε, υλοποίησης της νέα αγοράς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς θα οργανωθεί αυτή η νέα αγορά στο μέλλον αν δεν ξέρουμε και δεν ακούσουμε ποιες είναι οι προθέσεις της Επιτροπής για τη μελλοντική οργάνωση της αγοράς. Ευχαριστώ Ντένις. Πασκάλ Λεμπό. Ευχαριστώ. Βίκυ, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα σε αυτά που μόλις ακούστηκαν και που ανακοινώθηκαν σαφέστατα για το θέμα του TTIP και τις δυνατότητες που έχει ακόμα το Κοινοβούλιο να δράσει σε κάποια ζητήματα. Θα ήθελα καταρχάς και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έργο της. Θεωρώ ότι πραγματικά υπάρχει διάθεση να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις των ΜΕΝ και των ΔΕ και χαίρομαι γι' αυτό. Ε, το φορολογικό ζήτημα όμως ε, και τις παρατηρήσεις για τη φορολογική εναρμόνιση ε, είναι ένα από τα θέματα για τα οποία καταθέσαμε τροπολογίες. Εγώ δεν θα έθετα την ίδια στάση πολιτικής σύγκρουσης μεταξύ μας. Ναι, βέβαια, μπορεί να υπάρξει συζήτηση από αυτόν, αλλά αν ε, κατάλαβα καλά από την ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ, διότι ήρθε δύο φορές εδώ ενώπιον του Κοινοβουλίου, ε, είπε ότι αρχίζει να γίνεται ένα από τα ε, πιο σημαντικά θέματα της πολιτικής συζήτησης και της απαραίτητης εφαρμογής μιας Ευρώπης που θα συγκλίνει περισσότερο στα ζητήματα αυτά γεγονός το οποίο θα μας επιτρέψει να βρούμε τη χρηματοδότηση που χρειαζόμαστε για να υπάρξει βοήθεια για να τις επενδύσεις και να τα συνδυάσουμε και με τις ιδιωτικές επενδύσεις που περιμένουμε. Εγώ δεν θα ήθελα λοιπόν να το διαγράψουμε έτσι τόσο γρήγορα με την ε, ε, αιτιολογία ότι μπορεί να δημιουργήσει ε, συγκρούσεις το φορολογικό ζήτημα, διότι είμαι πεπισμένος ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία τα οποία θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να μπορέσουμε μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτές τις δημόσιες πολιτικές. Ένα αυτό λοιπόν και επομένω είμαι ε, διατεθειμένος να ξανασυζητήσουμε τα θέματα αυτά με ρεαλιστικό τρόπο και όχι με πολιτικό τρόπο. Ε, αν και για μένα δεν θα ήταν και πρόβλημα να συζητήσουμε ε, πολιτικά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ε, τα υπόλοιπα σημεία τώρα δεν θα τα ε, συζητήσω με λεπτομέρεια, δεν θα σταθώ με λεπτομέρεια στις τροπολογίες μου, αλλά ε, να πω ότι τα κριτήρια της ε, Ευρώπης 2020 θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα. Η αγορά δεν θα πρέπει να είναι μια τυχαία αγορά και υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία βασίζονται στην βιώσιμη ανάπτυξη και είναι πάρα πολύ καλό να τα υπενθυμίζουμε, καθώς επίσης είναι καλό να υπενθυμίσουμε και την ανάγκη να γίνονται σεβαστές κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις, ε, κάποια περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, διότι έτσι θα μπορέσουμε να προασπίσουμε και τις αξίες ε, οι οποίες βοήθησαν να οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα πρέπει να χαθούν ε, με τη διάθεση αυτή να πηγαίνουμε πάντα προς περισσότερη αποτελεσματικότητα και περισσότερη ανταγωνιστικότητα. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει καμία ανάπτυξη και καμία βιώσιμη ανάπτυξη όταν είμαστε αντίθετοι σε ε, έννοιες οι οποίες είναι αλληλένδετες όπως είναι η αποτελεσματικότητα και ε, η ανταγωνιστικότητα. Ε, αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές. Μετά υπάρχουν κάποια πράγματα ε, στις λεπτομέρειες για την προστασία των κατανολητών, ε, τις συλλογικέ δράσεις, τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να έχει μια πολύ πιο στεναρή δράση και θα μπορούσαμε αυτό να το επενθυμίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το να είμαστε δυναμικοί, εξαιρετικό. Η κυρία Κραπίνη είναι στον κατάλογό μου. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο να μιλήσει. Να μου το πείτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές. Πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη έκθεση, πάρα πολύ σημαντική για μας και η λειτουργία της ενιαίας αγοράς περιλαμβάνει τα πάντα. Αν η έκθεση αυτή είναι κατάλληλα διατυπωμένη και με καλές τροπολογίες, όπως είπε και η συγγητρία, είμαι βέβαιη ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας ε, θέσεις. Εμείς βρισκόμαστε εδώ, διότι θέλουμε να έχουμε καλύτερη νομοθεσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ενία αγορά. Εγώ δεν είμαι σκιώδης εισηγήτρια, κύριε εισηγήτρια, είμαι απλώς μέλος της Επιτροπής και Προσπαθώ να είμαι παντού, να κρατάω ε, τα μάτια μου και τα αυτιά μου ανοιχτά και να παρακολουθώ τι γίνεται. Είναι η πρώτη μου θητεία και ε, ίσως χρειάζομαι περισσότερο χρόνο να καταλάβω κάποια πράγματα. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια πράγματα που άκουσα από την εισηγήτρια. Θα μπορούσατε να μου πείτε για παράδειγμα γιατί ε, η τροπολογία για τις ε, συστάσεις αναχώρα δεν σας βρίσκει σύμφωνη. Μήπως δεν κατάλαβα καλά. Ε, υπάρχει μια τροπολογία που λέει ότι οι συστάσει αναχώρα θα πρέπει να υποβάλλονται και στα Εθνικά Κοινοβούλια πριν από το Συμβούλιο. Και εσείς λέτε ότι δεν ε, ε, είστε απόλυτα σύμφωνοι με αυτή την, έκθεση, την τροπολογία. Ίσως δεν κατάλαβα καλά. Αλλά αν αυτό εννοείτε ότι δεν συμφωνείτε, ε, μήπως μπορείτε να με εξηγήσετε γιατί. Εγώ έχω διατελέσει υπουργό και ήμουνα και μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου της χώρας μου και προκειμένου να υποβληθεί μια έκθεση στο Συμβούλιο πρέπει να έχει γίνει δεκτή και από το πιο αντιπροσωπευτικό θεσμικό όργανο που είναι το Κοινοβούλιο και όχι η κυβέρνηση. Βεβαίως το πότε θα πρέπει να γίνει η όλη διαδικασία είναι άλλη υπόθεση, αλλά είναι πολύ καλό να συμμετέχουν και τα εθνικά κοινοβούλια. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να συμμετέχουμε και ζητήσαμε από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας αντιμετωπίζουν επίσης όρις και να έχουμε κι εμείς λόγο από αυτό. Γιατί λοιπόν να μην συμμετέχουν και τα εθνικά κοινοβούλια. Επίσης, για την επανεβιομηχάνεια. Εσύ συμφωνώ με τον συνάδελφο που μίλησε προηγουμένως. Και πρέπει να σας πω το εξής. Πριν έρθω εδώ, ε, άκουγα συνεχώς ότι η Ευρώπη ε, χάνει τη βιομηχανία της. Και αν χάνουμε τη βιομηχανία μας πρέπει κάποιος να βρούμε έναν τρόπο να την ξαναποκτήσουμε. Και αν δεν το πούμε σε αυτή την έκθεση, πού θα το πούμε, αν δεν το πούμε στην έκθεση για την ενή αγορά. Ίσως χρειαζόμαστε μια διαφορετική διατύπωση, αλλά εξ όσων με αφορά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια αναφορά στην επανεκβιομηχάνηση. Ε, να σας ευχαριστήσω τώρα και ήταν πάρα πολύ δύσκολη η εκθεσή σας. Καταλαβαίνω ότι κάνετε πολύ σκληρή δουλειά. Ευχαριστώ να συγχαρώ κι εγώ με τη σειρά μου την εισηγήτρια για το έργο της. Θεωρώ ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και θα ήθελα απλώς πολύ σύντομα να συνοψίσω δύο ιδέες ε, από κάποια σημεία τα οποία παρουσιάστηκαν ε, προηγουμένως. Για να υπάρχει ε, στο εξάμεινο η σημασία και αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς για το, Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να προωθήσουμε δύο ειδώς. Καταρχάς να υπάρχει καλή νομοθεσία, η οποία όμως δεν αρκεί, θα πρέπει να είναι αποτελεσματική. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη η αποτελεσματικότητά της και θεωρώ ότι επειδή αρκετοί από εσά αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό και αναφερθήκαμε και στην ψηφιακή αγορά, όσο πιο ψηφιακή γίνεται ε, η αγορά μας, τόσο ε, λιγότερο εμφανής είναι η αποτελεσματικότητα. Είναι αντίστροφα. Η ψηφιακή αγορά είναι πάρα πολύ καλή, αλλά αναταράσει, διαταράσει τα πάντα. Επομένως, ε, στο θέμα αυτό των δικαιωμάτων, τα πάντα τα οποία διαταράσσονται από την ψηφιακή αγορά, θα βρεθούν ε, μπροστά μας οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, θα ε, μπορέσουν να αντιδράσουν πιο γρήγορα, αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι πιο ευάλωτες, αλλά η ενιαία αγορά εξαρτάται κατ' ουσίαν από τους οικονομικούς φορές, όπου έχουμε και τις μικρές επιχειρήσεις και φυσικά υπάρχουν και οι καταναλωτές εδώ και πρέπει να τους λάβουμε και αυτούς υπόψη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. οποιαδήποτε στοιχεία της ενιαίας αγοράς δεν έχουμε εκμεταλλευτεί, θα πρέπει να τα αναλύσουμε και να ε, διατηρήσουμε όλους τους καταναλωτές. Όταν θα δούμε λοιπόν τους δείκτες, θα πρέπει να περιλάβουμε όλους τους φορείς, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ε, αποτελεσματικότητα και επειδή αυτό είναι και έργο της Επιτροπές μας ε, και μας απασχόλησε και στην προηγούμενη θητεία, θα πρέπει να δούμε και τα δικαιώματα προσφυγής σε περίπτωση που δεν γίνονται σεβαστές οι διαδικασίες και η νομοθεσία. Ε, σε αυτά νομίζω ότι συμφωνούμε, γι' αυτό και είμαι πεμπισμένος ότι θα υπάρξει κάποια σύγκληση με τις κατάλληλες τροπολογίες, ε, συμβαστικές τροπολογίες. So, um, I don't see any other speakers. Does αν δεν έχουμε άλλους ομιλητές, η συγγετρία να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ζητήσω από την Επιτροπή να απαντήσει στην ερώτησή μου για το ότι η κοινοτική έκθεση στην εσωτερική αγορά δεν προσαρτήθηκε στις εκθέσεις των, ε, της εθνικές. Ο κύριος Τόγκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύντομα, πριν απαντήσω στην ερώτηση που μου τέθηκε, να πω σύντομα ότι χαιρετίζει η Επιτροπή το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής και την ε, σημασία που προσδίδει στην ενιαία εσωτερική αγορά και στο πόσο σοβαρά παίρνουμε το γεγονό ότι πρέπει να εμβαθύνουμε στην ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Ακόμη η έκθεση 2015 δεν έχει δημοσιευτεί και θα πρέπει να σας πω ότι εστιαζόμαστε εδώ στους τομείς που πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη σημασία. Όπως και εσείς, συμπίπτουν οι προτεραιότητες μας. Θα σας δώσω ως παράδειγμα την ψηφιακή ε, εσωτερική αγορά. Τώρα, και η εφαρμογή η σωστή είναι σημαντική και όχι μόνο οι παραβιάσεις. Θα πρέπει να ξέρουν διάφορε επιχειρήσεις ποια είναι τα δικαιώματά τους και πώς θα μπορέσουμε με ε, τα ψηφιακά μέσα να διευκολύνουμε την ολοκλήρωση αυτής της αγοράς. Η ψηφιακή τεχνολογία δεν είναι πάντα τροχοπέδι, αλλά και ένα πλεονέκτημα για τις μίμιες στην ενιαία εσωτερική αγορά. Τώρα, όσον αφορά το θέμα ε, που μου τέθηκε, δεν νομίζω ότι η Επιτροπή θεωρεί το γεγονό ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αναφορά στην ε, έκθεσή της έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους μας. Αν δείτε την ε, ετήσια έκθεση σε σχέση με τις προηγούμενες θα δείτε ότι προσδίδεται μεγαλύτερη σημασία στη ενιαία εσωτερική αγορά από ό,τι παρελθόν. Λέμε τι θα πρέπει να γίνει και σε κοινοτικό επίπεδο και σε εθνικό. Υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, αναλύονται οι αδυναμίες και τα προβλήματα και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δίδονται και στοιχεία ώστε να μπορέσουν οι διάφορες συστάσεις από το κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σωστά. Πιστεύω λοιπόν δεν θα πρέπει να το δείτε αυτό ως ενδιαφέρον ε, η, θέμα υποδέστερης σημασίας για την Κομισιό. Η νέα Επιτροπή αποφάσισε αυτή τη φορά να μην συμπεριλάβει την αναφορά στην οποία, την οποία εσείς μιλάτε, δεδομένου ότι έχουμε διαφορετικά μέσα αναφοράς για το θέμα αυτό. Έχουμε το scoreboard, έχουμε διάφορες εκθέσεις για τον τρόπο λειτουργίας της ενιαίας συνταγής αγοράς. Και θα πρέπει να θεωρήσουμε τα μέσα που έχουμε ώστε να καταλήξουμε σε κάτι το πιο αποτελεσματικό από ό,τι μέχρι σήμερα. Το επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε το 2015 το συντομότερο δυνατό στις αρχές του έτου να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε ένα στοιχείο αναφοράς, ένα μέσο αναφοράς που θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Δεν πάτε λίγο πιο αργά, σας προλαβαίνει και διερμηνείς, λέει πρόεδρος. Δεν είναι λοιπόν θέμα ε, σημασία στην οποία προσδίδουμε, επαναλαμβάνει ο εκπρόσωπο της Κομισιό, αλλά προσπαθούμε να βρούμε έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο αναφοράς αυτών των θεμάτων που αφορούν την ενιαία ιστορική αγορά. Εσύ γιατρία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ευχαριστώ για την εξήγηση, αλλά δεν με χαροποιεί και δεν ε, μου προσφέρει και νέα στοιχεία. Εάν είναι κάτι που θεωρεί η Κομισιό ότι είναι σημαντικό, δεν θα πρέπει να το παραγνωρίζει. Θα πρέπει μάλλον να τονίσει τη σημασία του. Θα τονίσει. Κανείς σημασία λέγοντας ότι του χρόνου θα σκεφτεί ένα καλύτερο μέσο παρουσίασης, μας κάνει να σκεφτόμαστε πολλά πράγματα σε ένα θέμα προσδίδουμε σημασία, του δίδουμε και προτεραιότητα και θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στην έκθεση που αφορά την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να είναι αυταπόδεικτο αυτό, να φαίνεται. Και θα πρέπει αυτό να το αναφέρουμε χωριστά και όχι να ζητούμε στους αναγνώστες να διαβάζουν ανάμεσα στις γραμμές. Η... οποία είναι σημαντικό θέμα και είναι πιο σημαντική από το ποσοστά μεταφοράς κοινωτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο της κάθε χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας. Ευχαριστώ τους συγγετή και τους συναδέλφους. Συμφωνώ με τα περισσότερα σχόλια που έγιναν και όπως προανέφερα είμαι στην ευτυχή θέση η μεγάλη πλειοψηφία των τροπολογιών να πω ότι ευθυγραμμίζονται με το περιεχόμενο της έκθεσής μου και της απόψης μου, άρα εύκολα θα καταλήξω σε συνενετικές διατυπώσεις και θα σας παρουσιάσω μια συνενετική έκθεση. Ίσως υπάρχουν και κάποιες ε, παρανοήσεις για κάποια θέματα. Εγώ δεν μπόρεσα να τα εξηγήσω σωστά. Όσον αφορά την τροπολογία του κύριου Γκουάγκας, συμφωνούμε με το μεγαλύτερο μέλος και το ίδιο ισχύει για την κυρία Γκρατίνη. Τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να επομιστούν τις ευθύνες τους. Θέλουμε να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία αλλά κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων μας και το επαναλάβω, βάνουμε συχνά, έχουμε την εντύπωση ότι δεν έχουν την εντύπωση πολλές φορές ότι κάποια πράγματα γίνονται εν τη απουσία τους και δεν τα αφορούν. Θα πρέπει όμως να συμμετέχουν πιο ενεργά σε όλη την διαδικασία αυτή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς θέλουμε τουλάχιστον στο δικό μας τομέα να το προωθήσουμε όσον αφορά τις τριμηνιές εκθέσεις. Οι τριμηνιές εκθέσεις υποβάλλονται σε μικρά χρονικά διαστήματα, όπως ξέρετε, και ίσως πολλές φορές δεν δίδεται χρόνος από τη μία έκθεση στην άλλη να έχουμε όλα τα στοιχεία τα οποία θέλουμε, ακόμη και στα ε, με την χρησιμοποίηση των ε, νέων ε, τεχνολογικών μέσων ώστε να συμπεριλαμβάνονται κάθε φορά στην έκθεση. Νομίζω ότι η στην κομισιόν της εκθέσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται και οι διάφορες συστάσεις που γίνονται στις χώρες θα το παρουσιάσω σωστά το θέμα αυτό, αλλά εν είμαι και ανοιχτή σε περαιτέρω τροπολογίες. Επίσης, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία αφορούν ε, την ε, φορολογική πολιτική και τις ε, ενέργειες κάποιων αποφύγουν την φορολογία. Νομίζω όμως ότι εδώ υπησέρχεται πολύ το πολιτικό στοιχείο θα προσπαθήσω να το εκφράσω σωστά το θέμα. Συμφωνώ με τον κύριο Ρόκφορτ, θα πρέπει η νομοθεσία να είναι και καλή στη θεωρία και αποτελεσματική. Στον τομέα των υπηρεσιών και των αγαθών θα πρέπει η νομοθεσία να είναι κατάλληλη ώστε τα προβλήματα που υπάρχουν και τα κενά στην ενιαία εσωτερική αγορά να ξεπεραστούν σιγά σιγά. Και πάλι θα ήθελα να παρακαλέσω την Επιτροπή να ξαναεξετάσει την προστασή της και να ζητήσω από τους σκιώδεις εισηγητές να υιοθετήσουν μία ενιαία θέση ώστε ή να κάνουμε μία ε, που βάλουμε ένα ενιαίο ερώτημα στην Κομισιό ή μία κοινή τροπολογία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρο και θα κάνω την συνενετική έκθεση. Ευχαριστώ. Θα έπρεπε να πω ότι είπα σήμερα, θα επαναλαβώ ότι είπα σήμερα το πρωί στη συνεδρία, λέει η Πρόεδρος. Δηλαδή, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ε, των ε, Επιτρόπων και της ε, διάσκεψης των Προέδρων που έγινε χθε το βράδυ και στην οποία συμμετείχα εξ ονόματος της Επιτροπής μας. Ο κύριος Κατάινεν υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να εμβαθύνουμε τη λειτουργία της ε, ενιαίας εσωτερικής αγοράς και στις ε, δράσεις μας για την σωστή εφαρμογή όλων των κανόνων. Είπα και Επιτροπής μας ότι εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι στα πλαίσια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν άκουσα όμως κανένα σχόλιο εκ μέρους του Επιτρόπου. Θέλουμε όντως να εφαρμοστεί σωστά η πολιτική με την οποία ασχολούμεθα, αλλά με ποιο τρόπο, πώς προτίθεστε να το κάνετε αυτό, με πιο αποτελεσματικά. Και σήμερα το πρωί, σήμερα, σε μία από τις πρώτες μου παρατηρήσεις, είπα ότι το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε με τους συντονιστές για να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε εμείς ε, να παρακολουθούμε και να υποπτεύουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό, δηλαδή η εμβάθυνση της ε, ενιαίας εσωτερικής αγοράς και η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων που πρέπει να ισχύουν. Και θα συζητήσω με τους συντονιστές αργότερα, γιατί θα επανέλθω στο θέμα αυτό και θα δούμε σε τι συμπέρασμα θα καταλήξουμε. Θα αλλάξουμε θέση, γιατί είμαι η εισηγήτρια για την επόμενη έκθεση και η κυρία Στάιλερ θα προεδρεύσει. Και καλύτερα να μην προεδρεύω ώστε να ακούσω τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι για την δική μου έκθεση. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε λοιπόν την Πρόεδρο να μας παρουσιάζει την έκθεση για την οποία είναι αρμόδια. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση λοιπόν, να ακούσουμε την έκθεση για την, ε, τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Η Βίκη Φόρντ είναι λοιπόν ε, αρμόδια. Ε, να ακούσουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν μιλήσει η, η συγγήτρια. Παρακαλώ, Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Γεια σας, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε συνοπτικά την ε, εκτίμηση επιπτώσεων για τα ατομικά μέσα προστασίας Αναθέσαμε δύο εξωτερικές μελέτες για το θέμα αυτό, καθώς και μία δημόσια διαβούλευση και θα ήθελα να πω ότι 77 απαντήσεις πήραμε στη δημόσια διαβούλευση 18% από τον, 27% από τον ιδιωτικό τομέα, 18% από το δημόσιο και άλλα ποσοστά από ε, κοινοποιημένα όργανα, από όργανα τυποποίησης και από ιδιώτες. Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, αν θέλετε όλες αυτές τις λεπτομέρειες μπορώ να σας τη στείλω 27% λοιπόν των απαντήσεων μας δόθηκαν από επιχειρήσει, 18% από τις ε, βιομηχανικές ομοσπονδίες, 22% με συγχωρείτε, 21% λέει ο μιλητή από ιδιώτες, 14% από εθνικές αρχές και 20% από κοινοποιημένους οργανισμούς και οργανισμούς τυποποίησης. Κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας συζητήθηκαν διάφορα θέματα στα πλαίσια της ε, ειδική ομάδας εργασίας με εκπροσώπους των κρατών μελών, των καταναλωτών, εκπροσώπων των οργανισμών τυποποίησης και των κοινοποιημένων οργανισμών. Η πρόταση ήταν, η πρόταση τελικά έγινε αποδεκτή φέτος στις 27 Μαρτίου. Τα κύρια θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε κατά την διάρκεια της ε, ε, εκτίμησης επιπτώσεων ήταν πώς θα γίνει ευθυγράμμιση με το παρόν ε, νινιπή, ποιο θα είναι το νομικό μέσον, η νομική βάση που θα ισχύσουν. Αν αφορά την ευθυγράμμιση, πρόκειται για μια διαθεσμική δέσμευση Στην αναθεώρηση της νέας νομοθεσίας θα πρέπει να μπορέσουμε να ευθυγραμμιστούμε με το νέο NINIP. Και θα δούμε ποιες είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε να μπορέσουμε να ενεργούμε σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μην υπάρχει δυσκολία και να μην υπάρχει υπερβολικό άχθος για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή για τα κοινοποιημένα όργανα. Όταν κάναμε αξιολόγηση της ε, κάλυψης, μάλλον δεν κάναμε τέτοιου είδους κάλυψη, δεδομένου ότι κάθε χώρα ενεργούσε διαφορετικά Υπήρχαν διάφορες εξαιρέσεις που αφορούσαν τα γάντια, που φορούν με στον οικοκυριό και ζητήθηκε ευθυγράμμιση για το θέμα αυτό, διότι για 25 χρόνια καλύπτονται από την ίδια οδηγία τα γάντια που φοράει κανεί για επαγγελματικούς λόγους, προστασία τα γάντια για ιδιωτικού λόγους και δεν μπορεί να καλυφθούν και τα δύο ήδη αυτά από την ίδια οδηγία. Δεν μπορούν να απολούνται χωρίς καμία διαφοροποίηση στα σούπερ μάρκετ. Είχαμε προβλήματα με άλλα προϊόντα. Όσον αφορά επίσης τις στατιστικές για ατυχήματα. Προσπαθήσαμε να εξετάσουμε αυτές τις στατιστικές, αλλά δεν συλλέγονται από τα κράτη-μέλη, άρα επισήμως δεν υπάρχουν και προσπαθήσαμε να ζητήσουμε από τα κράτη μέλη να μας δώσουν στοιχεία. Μας έδωσαν κάποια γενικά στοιχεία, αλλά αν... πολλές φορές δεν είχαμε περαιτέρω στοιχεία εάν καταστρεφόταν το προϊόν, αν το ανέφεραν οι ιδιώτες. Επίσης, όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα φορώντας τέτοιου είδους ε, γάντια. Δεν είχαμε σαφή ιδέα. Δεν ξέραμε ότι σε κάθε περίπτωση φορούσε κανεί, είχε κανείς την κατάλληλη ατομική προστασία. Κατά τη διάρκεια της εκτίμησης επιπτώσεων ζητήσαμε από τους εκπροσώπους των κατασκευαστών αν με τα προϊόντα αυτά υπάρχει πρόβλημα. Και οι απαντήσεις τους ήταν ότι δεν υπήρχε πρόβλημα. Διότι όσοι κατασκευαστές ε, κατασκεύονταν αυτά τα προϊόντα, διατείνονταν ότι παρέχουν και την κατάλληλη προστασία, χωρίς συμπληρωματικό κόστος. Παρ' όλα αυτά, όταν έχετε κατασκευαστές που προτείνουν προϊόντα προστασίας και από τεχνικής πλευράς δεν προστατεύει το προϊόν το οποίο κατασκευάζουν. Θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι αυξάνεται το κόστος κατά 10 με 20%. Ούτως ή άλλως ό,τι και να γίνει, πρέπει τα προϊόντα αυτά, να είναι προϊόντα προστασίας, να προσφέρουν προστασία. Η αγορά της, των ε, γαντιών κυρίως είναι αγορά στην οποία εξαρτώμεθα από εισαγωγής, αλλά δεν έχουμε επιμέρους στοιχεία. Πρόκειται όμως για αγορά 1,5 δις και η κοινοτική αγορά στον τομέα αυτό το κοινοτικό μερίδιο είναι 100.000 ευρώ μόνο. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τα γάντια για τον κήπο, τα προστατευτικά ή τον, τα γάντια που φορούν οι νοικοκυρέ για να κάνουν τι δουλειέ του. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε πάλι προϊόντα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύσουν τον χρήστη τους, αλλά βλέπουμε ότι δεν ακολουθούνται πάντα οι κατάλληλες διαδικασίες και όταν γίνονται οι μελέτες και οι έρευνες δεν είναι πάντα ο χρήστης προστατευμένος. Τι όσον αφορά την έκθεση σε υπερβολικό θόρυβο. Έχουμε ένα πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό. Ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να φορούν ειδικά ακουστικά προστασίας οι χρήστες, αυτοί που εκτίθενται σε τέτοιου είδους θόρυβο, τον οποίο πάνω από ένα επίπεδο θεωρούμε ενοχλητικό. Αφορούν τασπίδες, Φερρυπίν. Μιλούμε εδώ για προϊόντα της κατηγορίας 3. Και εκτός από τον κατάλληλο σχεδιασμό θα πρέπει τα προϊόντα αυτά να προσφέρουν υψηλό βαθμό προστασίας. Οι αμερικάνικες εταιρείες γενικότητα έχουν ένα σύστημα καλύτερης προστασίας και προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια. Ενώ τα προϊόντα τους είναι και πιο φτηνά. Εάν δεν έχουμε καλή ποιότητα ευθύς εξ αρχής για να βελτιωθεί η ποιότητα και η προστασία προσφέρουν τέτοιου είδους προϊόντα θα πρέπει να προβλέψουμε ότι αυξάνεται και το κόστος. At Επίσης υπάρχουν τρία τεχνικά κριτήρια στα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται ο κατασκευαστής. Και αυτό που μάθαμε από την εφαρμογή της σχετικής οδηγίας είναι ότι αυτά τα τρία τεχνικά κριτήρια δεν προσφέρουν καμία χρησιμότητα στον χρήστη. Είπαμε λοιπόν ότι καλύτερα να τα αποσύρουμε ώστε να μειωθεί και το κόστος για τον κατασκευαστή και για το κοινοποιημένο όργανο το οποίο δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με τόσο πολύπλοκα από τεχνικής πλευράς κείμενα. Δεδομένου ότι πρόκειται για κριτήρια πολύπλοκα από τεχνικής πλευράς. Τελικά, η αλλαγή της οδηγίας σε κανονισμό, κατά πρώτο λόγο για τους κατασκευαστές είναι διευκόλυνση, δεδομένου ότι δεν έχουν να κάνουν με 28 διαφορετικά κείμενα, αλλά με ένα ενιαίο κείμενο στη διάθεσή τους όλες τις κοινοτικές γλώσσες. Σε σχέση με την αρχή της επικουρικότητας, επίσης, είδαμε ότι στον κανονισμό υπάρχουν τεχνικά ε, προδιαγραφές και διατάξεις που πρέπει να είναι οι ίδιες σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πρέπει οι απαιτήσει και οι κανόνες να είναι οι ίδιες για όλους. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τεχνικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν όταν μεταφερθεί ο κανονισμός στην Εθνική Νομοθεσία με τον ίδιο τρόπο για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω εξηγήσει σχόλια εκ μέρους του συναδέλφου σας, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή για αυτή την παρουσίαση της αξιολόγησης επιπτώσεων σας ευχαριστώ, λέει η συγκήτρια. Έχω πολλά ερωτήματα. Σας ευχαριστώ γιατί οι σκιώδεις μου έχουν βάλει ήδη κάποια σχόλια. Το θέμα της ασφάλειας, των προτύπων ασφαλείας, του εξοπλισμού όπως γυλαίκα, γάντια είναι πάρα πολύ σημαντικά και βεβαίως κάτι που θα κάνει αυτή η νομοθεσία είναι να σιγουρευτεί ότι οι εισαγωγή από άλλες χώρες αυτού του εξοπλισμού εκτός Ευρώπης θα πρέπει να ε, τηρούν τα ίδια πρότυπα που καλούνται να τηρήσουν οι κατασκευαστές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ερωτήσεις μου λοιπόν, στην δήλωση συμμόρφωσης αν κατάλαβα καλά στο παρελθόν, ο κατεσκευαστής έπρεπε απλώς να δηλώσει ότι συμμορφώνεται κτλ. Σήμερα όμως θα πρέπει το κάθε αντικείμενο, ακόμα και αντικείμενα πολύ χαμηλής αξίας, να ε, συνοδεύονται από ένα πιστοποιητικό και να υπάρχει έλεγχος. Το ερώτημα εδώ είναι αυτό είναι προαιρετικό και ποιο θα είναι το επιπλέον κόστος ιδιαίτερα για πολύ ε, ευτελή αντικείμενα. Στο παράρτημα 5 εδώ βλέπω ότι προτείνεται να υπάρχει έγκριση για τα τελευταία, μάλλον ε, ε, άδεια κοινοτική η οποία έχει ισχύει πενταετή και ότι μετά θα πρέπει να ξεκινήσει νέα διαδικασία από μέρους του κατασκευαστή. Αυτό καταλαβαίνω. Έχετε κατανοήσει ότι αυτή η πρόταση έχουν κάποιες συνέπειες και ποιες είναι αυτές. Έχετε κάνει εξελόγησή τους. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι εξοπλισμού που ουσιαστικά ε, έχουν μπει σε κατηγορίες ανάλογα με την σημασία τους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Κατηγορία 2, παραδείγματος χάριν, γυλαίκα, σωσίβια που σας προστατεύουν από τον πνιγμό, θα μπορούσαν να μπουν στην κατηγορία 3. Εδώ κατά κάποιο τρόπο υπονομεύουμε τα πρότυπα. Έχετε ε, κάποια εξήγηση γι' αυτό. για κάποια άλλα μέσα σωστικά σε σχέση πάντα με τα σωσίβια. Εδώ ίσως θα πρέπει να δούμε σε ποια κατηγορία τα κατανέμουμε γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονομεύσουμε την ε, κατάταξη αυτή. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τώρα. Αναφέρεστε σε 77 απαντήσεις, εκ των οποίων το 27% ανταποκρίθηκε. Μα εδώ μιλάμε για πάνω από 4.000 επιχειρήσεις που εμπλέκονται στον τομέα αυτό και κατασκευάζουν αυτά τα αντικείμενα. Δεν ξέρω. Κάποια στιγμή διαβάζω στο κείμενό σας ότι το κόστος είναι μηδαμινό, γιατί υπάρχει <clears throat> μαζική παραγωγή. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν κάποιες πολύ μικρές ε, επιχειρήσεις και κατά κάποιο τρόπο δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα. Μπορείτε να μας δώσετε την πραγματική ε, σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα αυτό, με αριθμούς. Επίσης, αναχώρα τα στοιχεία που αφορούν ε, τα εγκάβματα και εδώ υπάρχουν επίσης ε, κάποια στοιχεία τα οποία όμως δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς πώς τα κατανέμετε. Μιλήσατε επίσης και για τις απαντήσεις, τις αρνητικές, λέγοντας ότι 18 απαντήσεις ήταν κατά κάποιο τρόπο αντίθετες, γιατί αυτές οι 18 βαρύνουν περισσότερο από τις 13 που είχαν την αντίθετη άποψη. Μπορείτε να μου πείτε επίσης, επανέρχομαι πάλι στο κόστος, ποια ακριβώς αντικείμενα έχετε συμπεριλάβει και ποια είναι, ε, ποιος είναι ο υπολογισμός του κόστους ακριβώς που έχετε κάνει, του επιπλέον κόστους, για τα αντικείμενα αυτά, αν συμπεριληφθούν και αυτές οι επιπλέον προδιαγραφές. Τελευταίο ερώτημα. Νατολογική σκέψη 9. Αναφέρεστε στην εξαίρεση κάποιων προϊόντων όπως τα χειροποίητα γάντια, λέγοντας ότι αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται. Αυτό δεν το βλέπω πουθενά εγώ στο κείμενο. Στην προηγούμενη οδηγία τα αντικείμενα αυτά με πολύ ρητό και σαφή τρόπο εξαιρούνταν. Γιατί καταρχήν εξαιρείται αυτά τα προϊόντα. Καταρχήν τι σημαίνει χειροποίητο γάντι και γιατί υπάρχει στην ιτελογική σκέψη και όχι στο κείμενο αυτό καθεαυτό. Να πάρουν το λόγο τώρα οι συγητές. Καταρχήν ξεκινάμε με το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα γερμανικά. Νομίζω ότι θα συμφωνήσει το σύνολο των συναδέλφων ότι είναι πολύ λογική και καλή αυτή η πρόταση από τη στιγμή που υπάρχει καλύτερη προστασία, καλύτερη και περισσότερη ασφάλεια για όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν και οι εισαγωγείς και οι κατασκευαστές και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται και στην συνάντηση των σκιωδών εισηγητών θίξαμε κάποια σημεία. Θα τα απευθύνω εδώ. Υπάρχουν οι ερωτήσεις της εισηγήτριας, στις οποίες συμφωνούμε. Το θέμα των περιορισμών. Κάπου βλέπω εδώ, στο άρθρο 5, 6 παραγραφός 2 στο I και στο J σημεία το θέμα των πιστοποιητικών που έχουν διάρκεια πενταετή. Και το ερώτημα εδώ είναι αν παραδείγματο χάρη υπάρχει ένα πιστοποιητικό και δεν έχει αλλάξει τίποτα στο προϊόν στη διαδικασία χρήσης γιατί υπάρχει προθεσμία, γιατί πρέπει ο κατασκευαστής να πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου την διαδικασία αδειοδότησης. Ποιος είναι ο σκοπός αυτός πίσω από την πρόταση της Επιτροπής να θεσπίσει πενταετή χρονική περίοδο. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ ευτυχείς ε, οι κατασκευαστές με αυτή την πρόταση. Δεύτερο, το θέμα των ε, των ε, αντικειμένων που ουσιαστικά γίνονται κατά παραγγελία, που δεν παράγονται μαζικά ιδιαίτερα όταν υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος και υψηλός κίνδυνος. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι πώς θα μπορούμε να μετρήσουμε αν θέλετε τα αντικείμενα αυτά, τα προϊόντα αυτά και να τα θέσουμε στην κατηγορία που ανήκουν. Και αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με το βαθμό επικινδυνότητας. Οι κατηγορίες 1, 2, 3 αν θέλετε, έχουν ε, δημιουργηθεί βάσει του βαθμού επικινδυνότητας. Γιατί λοιπόν αυτομάτως μπαίνουν στην κατηγορία 2. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν είναι θέμα αξίας ή τιμής, είναι θέμα βαθμού επικινδυνότητας, επαναλαμβάνω. Στο άρθρο 8, παράγραφος 6, το θέμα δηλαδή των ε, ενδείξεων που θα πρέπει να βρίσκονται σε φύλλο χαρτί, τυπωμένα λέει εδώ η πρόταση, γιατί όχι με άλλο τρόπο να μπορεί να τις βρει στο ίντερνετ παραδείγματος χάρη. Άρθρο 2, άλλο σημείο. Τι ακριβώς εννοείται εδώ όταν λέτε... Δεν, δεν καταλαβαίνω όταν λέτε ότι θα πρέπει να αναγράφονται με εμφανή τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βέσφαλ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά θα μιλήσω ε, λίγο γιατί δεν έχω φωνή, έχω βραχνιάσει. Αν κατάλαβα καλά αυτό που είπε η Επιτροπή, το θέμα το οποίο ήδη βρίσκεται στον τύπο ήδη στην ε, Γερμανία για το θέμα των γαντιών που χρησιμοποιούνται από τις νοικοκυρές. Ξέρουμε ότι σήμερα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες που κατασκευάζουν αυτά τα γάντια και το θέμα των ε, εγκαυμάτων Κοιτάξτε, όλοι ξέρουμε, όλοι και στη Γερμανία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν εκεί που κάποιος νιώθει σίγουρος και ασφαλής, στο σπίτι του δηλαδή. Δύσκολα λοιπόν θα καταλάβει κάποιος αν παραδείγματο χάρη εδώ προτείνουμε κάτι τέτοιο και Ουσιαστικά σαν αποτέλεσμα θα έχουμε την αύξηση της αμφισβήτησης της Ευρώπης και του ευρωσκεπτικισμού, εάν ε, προτείνουμε τέτοια πράγματα. Τι να σας πω, εγώ μαγειρεύω πάρα πολύ στο σπίτι μου. Δεν είμαι η μόνη βεβαίως και καταλαβαίνετε ότι η θερμοκρασία ενός φούρνου είναι από 100 μέχρι 250. Εντάξει, αν ανοίξω το φούρνο και μου έρθει όλος ο ατμός ε, και καώ, αλλά δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση. Το θέμα είναι πώς θα πιάσω το ταψί που είναι μέσα στο φούρνο και θα το βγάλω έξι. Αν θα το κάνω με γυμνά χέρια ή προστατεύοντας τα χέρια μου. Τι να σας πω τώρα. Θεωρώ πραγματικά ότι η συζήτηση για αυτά τα θέματα είναι βεβαίως σοβαρή, απαραίτητη και λογική. Αλλά, αλλά οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως θα πρέπει να προστατεύονται. Αυτή είναι, αν θέλετε, και η δική μας αποστολή. Δεν αμφισβητώ λοιπόν την αποστολή μας. Και φυσικά δεν, αποστο... δεν αμφισβητώ εδώ ότι είναι αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προστατεύσουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Και φυσικά όταν μιλούσαμε για το ABS ε, και την αυτοκινητοβιομηχανία υποστήριξα τις προτάσεις της Επιτροπής. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε πού τοποθετείται η συζήτηση και να μην είμαστε υπερβολική στις προτάσεις μας, ιδιαίτερα όταν αυτό αυξάνει σημαντικά το κόστος αυτών των προϊόντων. Και στον τριμερή διάλογο το είδαμε αυτό, ότι βεβαίως τα συστήματα ABS και αερόσακη και άλλα προστατευτικά ε, αξεσουάρ αυτοκινήτων σαφώς και προστατεύουν τις ζωές των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να αποδείξουμε ότι η προστασία αξίζει την τιμή που προσδίδεται. Και αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ είναι ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για το οποίο αναφεράμαστε. Εγώ διάβασα στο γερμανικό τύπο ο υπουργό Οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας λέγοντας ότι έχει παρανοήσει η Επιτροπή για να μην ε, δημιουργήσουμε λοιπόν τέτοιες αντιδράσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σας παρακαλώ πολύ να θέσουμε συγκεκριμένα, αν θέλετε, μηνύματα στην ευρωπαϊκή συζήτηση και να μιλήσουμε για ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Επαναλαμβάνω, δυστυχώς δεν έχω πολύ φωνή. Δυσκολεύομαι να μιλήσω γι' αυτό, θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Έχω κάτι καραμέλες που στη τσάντα μου που μπορεί να σας βοηθήσουν. Θα σας τα δώσω μετά. Ο κύριος ε, Ροσφόρ. Ευχαριστώ. Πριν ε, ξεκινήσω να σχολιάζω την έκθεση, θα ήθελα να σας πω ένα δυσάρεστο νέο που μόλις έμαθα ο Ζακ Μπαρό, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, ε, μόλις απεβίωσε. Ήταν ε, ο Γάλλος ε, Ευρωπαίος Επίτροπος πριν από τον Μισελ Μπανιέ και είναι ιδιαίτερα λυπηρό αυτό για μένα, ίσως και για σας. Ήταν και φίλος προσωπικός αλλά και πολιτικός φίλος και προασπιστής των ευρωπαϊκών ιδεών. Συλληπιτήρια λοιπόν. Απεβίωσε στις 3 η ώρα στο μετρό στο Παρίσι. Υπάρχουν τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον, όσον αφορά τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, είμαι σε δυσάρεστη θέση, διότι αφενός νιώθουμε ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλά δεδομένα, αλλά ταυτόχρονα νιώθουμε ότι η διαβούλευση δεν ήταν ε, απόλυτα επίσημη και αυστηρή. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, ε, οι οποίες είναι ανεπαρκείς όμως. Επομένως εδώ υπάρχει ένα ερώτημα και φυσικά δημιουργούνται ερωτηματικά και για τις πιθανές επιπτώσεις το είπαν και οι συνάδελφοι άλλωστε, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά το θέμα της εκτίμησης των επιπτώσεων ε, δεν ε, είμαι κατά σε καμία περίπτωση και ε, δεν θέλω να νομίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή ζητάμε πιο συγκεκριμένε πληροφορίες για το θέμα αυτό αυτό σημαίνει ότι έχουμε επιφυλάξει ή είμαστε αντίθετοι στην πολιτική κίνηση που θα κάνουμε από αυτού ίσα ίσα εγώ το υποστηρίζω αυτό που θέλουμε να κάνουμε κυρίως στο θέμα των ατοχημάτων στο σπίτι, στην καθημερινότητά μας ότι η προστασία είναι ε, για ε, το, ε, την οικογενειακή μας ζωή, την καθημερινή μας ζωή υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα και μάλιστα είναι περισσότερα από τα τροχαία ατυχήματα. Ε, θα θέλαμε λοιπόν κάποια συμπληρωματικά στοιχεία από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το... Ε, κατά πόσον είναι απόλυτα αυστηρά τα όσα μας είπε στη διαβούλευση. Ε, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αντικειμένων, όντως ε, το είπατε κι εσείς. Ε, και ε, τα γάντια ε, της κουζίνας για να βγάζει ε, κάποιος το ταψί από το φούρνο δεν είναι αποκλειστικό αντικείμενο για τις γυναίκες για να σκεφτώ και λίγο και άντρες βγάζουν τα ταψιά του φαγητού από το φούρνο ε, ίσως επειδή εγώ είμαι σοσιαλιστής και είμαι αριστερός ε, ε, βρέθηκα ε, στο νοσοκομείο ακριβώς γιατί πιάνουν τα χέρια μου και βρέθηκαν να φαίνω διάφορα τυχήματα. Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι εύκολο να το ρυθμίσουμε. Για παράδειγμα, στη χώρα μου πολλά από αυτά τα γάντια είναι χειροποίητα και γίνονται στην επαρχία ή αλλού, έχουν και διάφορα τοπία επάνω. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ αυστηροί, διότι η θερμότητα μπορεί να μας χτυπήσει και αν ε, έχει καλό καιρό μπορεί να φάμε έξω στην πλατεία και να φέρουμε ένα πάρα πολύ ζεστό πιάτο και η αντίσταση στην ε, ε, θερμότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και υπάρχει και εξαίρεση, ναι, μεν υπάρχουν πράγματα χειροποίητα που κάνουν βιοτέχνε, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα. Εγώ δεν θέλω να καώ σε καμία περίπτωση. Θέλω να μπορώ να βγάλω το πιάτο μου, το ταψί μου από το φούρνο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ε, ε, είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητο στο επιχείρημα της ε, διαδικασίας, της επαχθούς και πραγματικά θεωρώ ότι τα επιχειρήματα του συναδέλφου από το ΕΛΚ όσον αφορά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ιστιακούς, διαδικτυακούς ιστότοπους για να δούμε τι θα κάνουμε μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο και τίθεται ερώτημα για το τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Δεν κατάφερα να βρω απαντήσεις ε, στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ερώτημα αυτό. Ε, η δυναμική του συστήματος. Εγώ πιστεύω και το συζητήσαμε και προηγουμένως με το θέμα του ε, περιορισμού της άδεια στα 5 έτη ότι καλό θα ήταν το σύστημα να είναι λίγο δυναμικό. Η ασφάλεια των προϊόντων δεν είναι κάτι δεδομένο, είναι κάτι το οποίο εξαρτάται πάρα πολύ από την έρευνα και από την ανάπτυξη, εξαρτάται από την καινοτομία και επομένω βρισκόμαστε ενώπιον μιας αντιφατικής κατάσταση και πάλι. Εάν υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός πάρα πολύ μεγάλος, αν είναι πολύ μεγάλη η διάρκεια, ε, ε, το να θεωρείται ένα προϊόν εξόψεως ασφαλές ε, θα βρεθούμε να υστερούμε ενώπιον των, της προόδου που γίνεται και το γεγονός ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την προστασία αυτών των προϊόντων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται, να βελτιώνεται, να λαμβάνουμε υπόψη νέα υλικά, νέες διαδικασίες επεξεργασίας ε, και όλα αυτά θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο να ε, είναι αρκετά ήπιο και ευέλικτο ώστε να μας επιτρέπει να μπορούμε να συμπεριλαμβάνουμε συνεχώς και νέες καινοτομίες. Τώρα, αν αυτό έχει σχέση με το συγκεκριμένο χρονικό όριο, δεν ξέρω. Αλλά ε, εδώ και η συζήτηση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντική και δεν είναι πάρα πολύ εύκολη, διότι αφενός βλέπουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς μπορεί να αυξηθεί το κόστος, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι και εξασφαλισμένες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το τι μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, για τις εισαγωγές, όπως είπε η Βίκυ Χόρτ προηγουμένω. Πρέπει να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι έχουν να αντιμετωπίσουν ε, έναν ανταγωνισμό ο οποίος πρέπει να είναι ισότιμος. Και εγώ θεωρώ ότι το να υπάρχουν επιπλέον ποιοτικά στοιχεία για να αυξηθεί η ασφάλεια θα πρέπει να έχει και ένα αντίτιμο. Αλλά το θέμα είναι ποια είναι η λογική τιμή. Πώς μπορούμε να καθορίσουμε τη λογική τιμή. Το να λέμε ότι το να συμπεριλάβουμε τα νέα στοιχεία που ενισχύουν την προστασία και την ασφάλεια των προϊόντων αυτών δεν ξέρω αν είναι πάντα δυνατόν. Ε, ο ανταγωνισμός θα πρέπει να φροντίσει να μην υπάρχει μεγάλη αύξηση των τιμών όταν πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές για να υπάρχει συμμόρφωση για κάποια νέα προϊόντα. Ε, όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν στο, αυτό, στο σημείο αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε επί της ουσίας, συμφωνούμε επί των κατευθυντηριών γραμμών, συμφωνούμε προς την ανάγκη να υπάρχει μία άμεση και μέγιστη εναρμόνιση στο μέτρο του δυνατού, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά τα οποία θα μπορούσαμε να τα θεωρούμε με λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι λεπτομέρειες στην πραγματικότητα, είναι θέματα ε, ε, οργανωτικά τα οποία θα πρέπει να σκεφτούμε και έχουμε πολλή δουλειά θεωρώ και με την εισηγήτρια για να μπορέσουμε να ε, έχουμε όσο το δυνατόν πιο εύστοχες απαντήσεις και αυτό θα κάνουμε σε επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστούμε κύριε Ροσφόρ. Ο κύριος Μαστάλκα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι καταρχήν οι περισσότερες ερωτήσεις που ήθελα να κάνω τέθηκαν από άλλους συναδέλφους. Το θέμα της θερμοκρασίας για να αποφευχθούν ε, τα ατυχήματα στο σπίτι. Εγώ εχθές είδα την παρουσίαση της Επιτροπής και είδα ότι υπάρχουν περίπου 4.000 επιχειρήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά που κατασκευάζουν αυτό τον εξοπλισμό. Και μόνο 77 συμμετείχαν. Είναι αρκετός ο αριθμός αυτών των επιχειρήσεων που συμμετείχε σε αυτή την αξιολόγηση. Έτσι ώστε να υπάρξει μια τέτοια τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αντιδράσουν εάν επιδεινωθεί η κατάσταση και γίνει πιο δύσκολη η διαδικασία ή πιο δαπανηρή. και πολλά στοιχεία που τους αφορούν σίγουρα δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν την αξιολόγηση. Θεωρώ λοιπόν ότι στα πλαίσια μιας τέτοιας μελέτης Σίγουρα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα στοιχεία από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι σημαντικοί παράγοντες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση για την Επιτροπή και να επανέλθω σε αυτά που είπε ο κύριος Οσφόρ για την σωστή τιμή για αποτελεσματικά προϊόντα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ορθό, έτσι όπως το έθεσε. Θα πρέπει δηλαδή να πληρώνουμε στη σωστή τους τιμή τα αντικείμενα αυτά. Δεν μπορούμε διαρκώς δηλαδή να λέμε ότι έχουμε καλύτερη ποιότητα και οι τιμές παραμένουν σταθερές. Κύριε Ροσφόρο, έχω κάτι να σας πω. Τι αγοράζουμε ποια είναι η τιμή του και πόσο χρόνο θα διαρκέσει το προϊόν αυτό. Ένας καταναλωτής, κατά την άποψή μου, είναι διατεθειμένος να πληρώσει ένα αντικείμενο για να μην κάψει τα χέρια του. Το θέμα είναι όμως πόσο διαρκεί το προϊόν αυτό, αν είναι ανθεκτικό. Και το θέμα της ασφάλειας τελικά βλέπουμε ότι είναι, έχει, είναι σε άμεση συνάρτηση με την διάρκεια ζωής του προϊόντος και της τιμής βεβαίως. Η ερώτησή μου τώρα προς την Επιτροπή. Συμφωνώ ότι όταν κάποιος κάνει μια ερώτηση μπορεί να ζητάει και πληροφορίες, δεν είναι απαραίτητο ότι διαφωνεί. Αναφερθήκατε στις τρεις απαιτήσει. Τις αναφέρατε και τις τρεις δονήσεις, μηχανικές κτλ. Είπατε με σαφή τρόπο ότι αν αυτές οι τρεις απαιτήσεις, τρία προαπαιτούμενα καταργηθούν, δεν θα έχει επιπτώσεις για τους εργαζομένους. Ερωτώ, ποια είναι τα κριτήρια στα οποία βασίζεστε, οι δηλώσεις των επιχειρήσεων ή έχετε και άλλα στοιχεία που στηρίζουν αυτή σας τη δήλωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. θα ήθελα να πω ότι εκπλήσωμαι πολύ ακούγοντας αυτή τη συζήτηση. Ουσιαστικά πρόκειται εδώ για μία πρόταση κανονισμού που δεν ξεκινάει από το μηδέν. Βασίζεται σε μία οδηγία του 89. Δηλαδή υπάρχει η βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε το νέο κείμενο. Δεν κάνουμε κάτι τελείως καινούριο. Αν κατάλαβα καλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θέλει ουσιαστικά να πλουστεύσει τις διαδικασίες και να κάνει ένα πιο κοινό κείμενο. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα ακούγοντας αυτό που προτείνει η Επιτροπή και θεωρώ ότι αυτή η αξιολόγηση αντικτύπου είναι πολύ σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πολλές ε, αξιολογήσεις επιπτώσεων, δεν είναι το πρώτο θέμα και είναι σημαντικό εδώ να υπάρξουν ερωτήματα και απαντήσεις. Βάσει αυτού, αυτής της διαδικασίας γίνεται και η αξιολόγηση αντικτύπου. Το θέμα λοιπόν είναι, αν θέλουμε να είμαστε λογικοί, να βελτιώσουμε την κατάσταση. Θέλω να κάνω μία παράκληση, μία έκκληση προς την γραμματεία της Επιτροπής. Δεν πρόλαβα να διαβάσω το κείμενο. Πολύ σύντομα το κοίταξα και θα ήθελα να μου πείτε, γιατί όταν προσπάθησα να διαβάσω τα παραρτήματα δεν βρήκα τίποτα. Δεν είχε κανένα κείμενο, τίποτα. Ούτε στο ίντερνετ, ούτε στο φάκελό μου. Γι' αυτό και πραγματικά επειδή με ενδιαφέρουν τα θέματα αυτά, το θέμα της ρήτρα Sunset παραδείγματο χάρη, κάτι που πάντα απέριψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν υπάρχει εδώ σε αυτό το κείμενο. Γι' αυτό και θα ήθελα να μου ξεκαθαρίσει η Επιτροπή ακριβώς τι συμβαίνει εδώ. Ξέρω ότι το Συμβούλιο έχει ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις του. Εμείς δεν έχουμε καν ξεκινήσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ρωτώ λοιπόν την εισηγήτρια ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και ούτε για τη δική σας έκθεση δεν έχουμε κάποιες ημερομηνίες και κάποιο χρονοδιάγραμμα. Μπορείτε να μας πείτε κάποια στοιχεία και για σας και για την, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Να δώσω το λόγο στην Επιτροπή αν συμφωνείτε. Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις και μετά θα δώσω το λόγο και στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επιτρέψτε μου καταρχήν να προσπαθήσω να αποσαφηνίσω την κατάσταση. Αν κατάλαβα καλά, υπάρχουν 4.000 επιχειρήσεις που παράγουν, κατασκευάζουν γάντια. Όχι, όχι για όλον τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας αναφέρεται αυτός ο αριθμός επιχειρήσεων. Πολύ λίγες παράγουν και κατασκευάζουν αυτά τα γάντια στην Ευρώπη και είναι συνήθως μικρές. Μικρές επιχειρήσεις που παράγουν, κατασκευάζουν αυτά τα γάντια για οικιακή χρήση. Για το φούρνο προστασία από θερμοκρασία. Λοιπόν, και όταν μιλήσαμε για τις 4.000 επιχειρήσεις αναφερόμασταν στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Επιχειρήσεων για αυτόν τον εξοπλισμό, για όλο τον εξοπλισμό, όλα τα προϊόντα. Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ζητήσαμε αν θέλετε, σε δύο διαφορετικές μελέτες. Είναι δημοσιευμένες, μπορείτε να τις διαβάσετε, είναι στη διάθεσή σας και υπάρχει αυτή η δημόσια διαβούλευση και τα αποτελέσματά της. Τώρα, για τα γάντια. Ποιος παρακολουθεί την αγορά, ποιες είναι οι αρχές εποπτείας της αγοράς. Αν θέλετε υπάρχουν παρόμοια γάντια με αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση, τα οποία αν θέλετε ε, έχουν ειδική σήμανση για επαγγελματική χρήση. Σήμερα ακόμα και τα γάντια για οικιακή χρήση, αν πραγματικά τηρούν τις προδιαγραφές οι κατασκευαστές, προστατεύουν και γι' αυτό και ο καταναλωτής τα αγοράζει. Ο κανονισμός αυτός δεν ζητάει περαιτέρω τεχνικές ε, προδιαγραφές και απαιτήσει. Τους λέει απλώς να τηρούν αυτό που λένε ότι κάνουν. Και αυτό ανταποκρίνεται και στο κόστος, αν θέλετε. Εδώ αναφερόμαστε σε μια αύξηση κόστου της του 10-20% που είναι το επιπλέον κόστος για τα γάντια αυτά που σήμερα δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το επίπεδο προστασίας όπως αναγράφεται και δηλώνει ο κατασκευαστής. Τα γάντια δηλαδή αυτά τα οποία παραδείγματο χάρη προστατεύουν και δεν προστατεύουν στην πράξη, αν αυτό το προϊόν έμπαινε στο πεδίο της, του κανονισμού, θα έπρεπε να αποσυρθούν από την αγορά. Σήμερα δεν γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί ακριβώς δεν καλύπτονται αυτά τα γάντια από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Και δεν μπορούμε να ζητήσουμε να αποσυρθούν από την αγορά. Αυτό είναι, περί αυτού πρόκειται και τίποτα παραπάνω. Τώρα, για τα άλλα θέματα. Το θέμα της πενταετίας και του, της πιστοποίησης. Ζητάμε ανανέωση. Δηλαδή, θα δοθεί ανανέωση αν δεν έχει αλλάξει το προϊόν και θα ζητηθεί νέο πιστοποιητικό αν έχει αλλάξει το προϊόν. Παραδείγματος χάρη για τα σωσίδια επειδή υπήρχαν προβλήματα με τη συμμόρφωση ζητήσαμε από ένα κατασκευαστή να τροποποιήσει το προϊόν και η απάντηση ενός ε, κατασκευαστή ήταν «Μα εγώ έχω πιστοποιητικό που ισχύει επάπειρον, άρα δεν έχω την υποχρέωση να αλλάξω τίποτα. Γι' αυτό μιλήσαμε για αυτήν την πέντα αιτία. Εάν τυχόν υπάρχει αλλαγή στο προϊόν, θα ζητηθεί νέο πιστοποιητικό, αλλιώς θα ανανεώνεται. Γι' αυτό και οι οργανισμοί πιστοποίησης θα πρέπει να συμπεριφέρονται ανάλογα με τα δεδομένα. Αν κάτι έχει αλλάξει θα υπάρξει εκ νέου εξέταση του προϊόντος και νέα πιστοποίηση, νέο πιστοποιητικό. Αν όχι θα ανανεώνεται το πιστοποιητικό. Και το κόστος δεν είναι σημαντικό σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, το θέμα των καταπαραγγελία προϊόντων, αυτών που κατασκευάζονται μετά από συγκεκριμένα αιτήματα. Γιατί μπαίνουν στην κατηγορία 2 αυτόματα αυτά τα προϊόντα. Γιατί. Στην κατηγορία 3 Ε, τα προϊόντα που βρίσκονται στην κατηγορία 3 περνάνε από μία διαδικασία παραγωγής. Αυτό δεν ισχύει, παραδείγματο χάρη, με το προϊόν που παραγγέλλεται επί τούτου και το οποίο κατασκευάζεται μία φορά με ειδική παραγγελία. Και αυτό και μπαίνει στην κατηγορία 2 γιατί δεν υπάρχει η διαδικασία μαζικής παραγωγής. Τώρα, δεν θεωρούμε ότι αυτό καθώς και το θέμα του επιπλέον κόστους θα πρέπει να συμπεριληφθεί κάπου αλλού στο κείμενο, υπάρχει στις αιτιολογικές σκέψεις. Τώρα, όσον αφορά, αν θέλετε, την απέτηση να υπάρχει σήμανση σε έγγραφη μορφή, αυτό δεν είναι τίποτα το καινούριο. Και όσον αφορά τη δυνατότητα να δοθούν οι πληροφορίες μέσω ίντερνετ, Σήμερα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση μία επιχείρηση να ανακοινώνει κάποια πράγματα στο ίντερνετ και αυτές οι πληροφορίες να παραμένουν πάντοτε προσβάσιμες στο ίντερνετ. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι πρέπει να ε, αναφέρονται πάνω στο προϊόν και με έγραφο τρόπο. Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι μηχανικές δονήσεις. Κοιτάξτε, αυτό μια γενική προϋπόθεση και προαπαιτούμενο. Οι μηχανικές αυτές δονήσεις θα πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με το κάθε ξεχωριστό εξοπλισμό προστασίας, γιατί το κάθε, ο κάθε εξοπλισμός έχει τελείως διαφορετική, διαφορετικό βαθμό προστασίας. Γιατί για κάποιον εργαζόμενο χρειάζεται γενική προστασία, αν όμως έχει ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό προστατευτικό, για, μια πολύ συγκεκριμένη, για ένα πολύ συγκεκριμένο μηχάνημα που προκαλεί πολύ συγκεκριμένες μηχανικές δονήσεις, Βεβαίως οι γενικές προδιαγραφές και τα προαπαιτούμενα ισχύουν, εδώ όμως θα πρέπει να προσθεθούν και κάποιες επιπλέον προδιαγραφές. Αυτό εννοούμε εδώ. Βεβαίως όλες αυτές οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις μελέτες μας ε, είναι στη διάθεσή σας, δεν υπάρχει θέμα. Μπορώ να σας ε, τροφοδοτήσω με όλες αυτές τις επιπλέον πληροφορίες και στοιχεία. Όλα τα στατιστικά στοιχεία και τα δεδομένα που έχουμε είναι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σύντομα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδελφούς ότι την έκθεση αυτή την επέλεξα εγώ διότι κανένας άλλος συνάδελφος ή ομάδα δεν την ήθελε. Και πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι είναι κάτι το εξαιρετικά ενδιαφέρον και για προσωπικούς λόγους την ανέλαβα και οποιαδήποτε άλλο σχόλιο με ε, πλητή βαθύτερα. Στην αρχή αρχίσαμε για τα θέματα προστασίας ε, ε, τομικής προστασίας όπως τα σωσίβια ή άλλα τα οποία είναι εξαιρετικά ε, σημαντικά και πιστεύω ότι στα πλαίσια του νέου νομοθετικού πλαισίου πρέπει να ισχύουν για όλους οι κανόνες. Υπάρχουν παρόλα αυτά ε, θέματα τα οποία στα πλαίσια όλων αυτών των δύο τα φίξαμε την προφορή στη συζήτηση. Εδώ έχουμε ε, παράταση του πεδίου εφαρμογής. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Θα πρέπει να δούμε εάν κάποια προϊόντα που αφορώνται στη συγκεκριμένη περίπτωση στην ίδια κατηγορία με κάποια άλλα ε, δεν αφορώνται. Και αν θέλουμε να έχουμε νέα νομοθεσία για τέτοιου προϊόντα, θα πρέπει να το κάνουμε με τρόπο να βοηθήσουμε τους κατανοητές και όχι να τους δημιουργήσουμε προσκόμματα. Ελπίζω ότι η έκθεσή μου και γι' αυτό το λόγο δεν έθεσα προθεσμία κατά στροπολογιών, γιατί θέλησα πρώτα απ' όλα να δω τους σχεδόν συζητητές και να συζητήσω μαζί τους. Χθε το βράδυ το έκανα Δυστυχώς δεν μπορούσε χθε το βράδυ να είναι παρούσα η συγγήτρια εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας γιατί έχει αναπρομία. Σε πάση περιπτώσει θα το διευθετήσω το θέμα. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 27 ε, Ιανουαρίου. Ίδια προθεσμία και για τις συσκευές αερίου. Θα πρέπει να δούμε αν κατά... Ε, ε, ευχαριστώ που διευκρινίσατε κάθε ε, κάποια σημεία όπως αυτό της πενταετούς διάρκειας. θα προσπαθήσω, αφού λάβω τις τροπολογίες και ηλεκτρονική ηλεκτρονική μορφή, να δω με απόλυτη σαφήνεια ποια είναι τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε αυτές τις κατηγορίες και βεβαίως τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε σε αυτή την περίπτωση, τα χρησιμοποιούμε τα γάντια συγκεκριμένα και για να προστατεύουμε γυναίκες στο μενικιούρ μας, αλλά κυρίως για να προστατεύουμε και τα χέρια μας από διάφορα χημικά βλαβερά προϊόντα. Είναι εξίσου σημαντικό. Πριν φτάσουμε στη τελική απόφαση, νομίζω ότι θα πρέπει να ξανασυναντηθούμε τους γητέ και να εξετάσουμε όλους τι τροποσίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία εισηγητρία και σας παραδίδω και πάλι την Προεδρία. Um, Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι εμπορικές πρακτικές ε, στον ε, τομέα ε, του, της διατροφικής αλυσίδας και να δώσω απευθείας το λόγο στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Um, yes. Ναι, σας ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Ιούλιο φέτος για τις ε, θεμητές εμπορικές πρακτικές ε, στον τομέα της διατροφικής αλυσίδας. Από ό,τι κατάλαβα τα μέλη θέλουν και κάποιες πληροφορίες για μια μελέτη που κάναμε όπου ζητήσαμε μία μελέτη για να εξετάσουμε την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Δεν θα τα κάνω ξεχωριστά. Στη διάρκεια της παρουσίασής μου θα συμπεριλάβω και κάποιες εξηγήσει για τον τρόπο με τον οποίο ε, έχει κατάσταση ε, στα κράτη-μέλη και αυτό είναι βάση της μελέτης. Πρόκειται για ένα ζήτημα όπου στην προηγούμενη θητεία υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον ε, από την Επιτροπή και ε, γενικότερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως για το λιανικό τομέα, που είναι και ε, τομέας βασικός για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Before we moving to, to the communication with a να ξεκινήσω λοιπόν με την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια σύντομη εξήγηση για το τι εννοούμε με τον όρο αθέμητε εμπορικές πρακτικές. Προσπαθούμε να ετοιμάσουμε έναν ορισμό. Πρόκειται για ε, πρακτικές οι οποίες παρεκκλίνουν από τις ε, καλές εμπορικές πρακτικές και ε, είναι αθέμητε. Παραδείγματο χάρη, κατάχρηση ε, ε, λόγω ασαφών ή ελλειπών πληροφοριών σε κάποια σύμβαση, ε, μονομερείς όροι ε, σε κάποιες συμβάσεις. Αυτή είναι μία από τις ε, ε, περιπτώσεις που αναφέρονται συχνά και τέλη ευνηδιαστικά τα οποία επιβάλλονται από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη μιας σύμβασης. Γιατί είναι προτεραιότητα το θέμα αυτό στη διάρκεια του τελευταίου έτους νομίζω ότι έχει σχέση με τα όσα συμβαίνουν στον τομέα της διατροφικής αλυσίδας. Στη διατροφική αλυσίδα υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, ελλείψεις ισορροπίας ε, λόγω διαπραγματευτικής δύναμης. Υπάρχουν μικροί και μεγάλοι παίκτες, ε, λίγοι μεγάλοι και μικροί player και από τις δύο πλευρές, παίκτες και από τις δύο πλευρές αγοράς και θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση του φαινομένου στη διατροφική αλυσίδα και αυτό φυσικά δεν ισχύει μόνο για το λιανικό τομέα, αλλά φυσικά και για κάποια πολύ σημαντικά προϊόντα ε, και για την πλευρά των προμηθειών. Έχουμε ε, ευμετάβλητες τιμές στις αγορές αγαθών, ε, πιέσεις των τιμών οι καταναλωτές έχουν σχετικά περιορισμένο προϋπολογισμό και δυστυχώς δεν μπορούν να καταβάλουν το αντίτιμο αυτών των προϊόντων και υπάρχει και ε, ε, αυξημένος κίνδυνος ακριβώς λόγω αυτού του γεγονότος για αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα προσφάτως. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει... Ε, μια εθελοντική ε, ε, πρωτοβουλία στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Σε επίπεδο κρατών μελών υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις. Υπάρχει ε, κάτι στο οποίο θα επανέλθω στην επόμενη διαφάνειά μου και σε επίπεδο κρατών μελών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε επίπεδο κρατών μελών έχουμε διάφορες αντιδράσεις. Υπάρχει νομοθεσία η οποία εισήχθε προκειμένου να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες αθέμητες εμπορικές πρακτικές, υπάρχουν κάποιες ε, αλλαγές ε, στο δίκαιο ανταγωνισμού ή και δίκαιο ανταγωνισμού το οποίο αφορά αθέμητες εμπορικέ πρακτικέ και εφαρμόστηκε γι' αυτό, παρόλο που δεν τροποποιήθηκε προσφάτω. Υπάρχουν και κάποια εθελοντικά προγράμματα πρόσφατα και υπάρχουν και κάποια κράτη-μέλη που δεν έχουν κάποιε συγκεκριμένε δράσει επί του θέματο. Η τάση όμω είναι να αυξάνονται οι πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών. Να σχολιάσω λίγο τώρα κάθε μία από αυτές τις πρωτοβουλίες λίγο πιο αναλυτικά. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταρχάς, Εδώ και κάποια χρόνια οι ενδιαφερόμενοι στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων έχουν ε, συμφωνήσει για ένα θελοντικό πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουμε τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Τελικώς υπήρξε συμφωνία ε, πριν από ένα χρόνο επ' αυτού. Και τώρα αποκαλείται η πρωτοβουλία αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους. Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει καταρχάς να επισημάνουμε ότι έχει μια σειρά αρχών και βέλτιστων πρακτικών και αυτές οι βέλτιστες πρακτικές έχουν συμφωνηθεί από όλους τους ενδιαφερομένους. Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο στη διαδικασία, το οποίο μας οδήγησε σε αυτή την πρωτοβουλία για την αλυσίδα εφηδιασμού τροφίμων. Ήταν μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι στην αλυσίδα ε, συμφώνησαν για μια σειρά από αρχές και βέλτιστες πρακτικές και υπάρχουν και παραδείγματα αυτών των βέλτιστων πρακτικών. Ωστόσο, τελικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι δεν προσυπογράφουν αυτή την πρωτοβουλία, κυρίως διότι υπήρξε απογοήτευση κάποιων εκ των ενδιαφερομένων λόγω των περιορισμών που είχε ε, σε, στην πτυχή της ε, συμμόρφωσης ε, η συμφωνία αυτή. Κάποιοι ενδιαφερόμενοι λοιπόν δεν κατάφεραν να προσυπογράψουν την πρωτοβουλία αυτή για την αλυσίδα εφοδιασμού του προφήμου... αλλά για τις αρχές συμφωνούν όλοι. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη τώρα. Σας ανέφερα ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία εισήγαγαν σχετική νομοθεσία που στοχεύει στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Τα βλέπετε τα κράτη-μέλη αυτά στο χάρτη. Υπάρχουν διάφορες λύσεις, είναι λίγο διαφορετικές. Ε, συνήθως υπάρχει ένας κατάλογος πρακτικών, απαριθμούμε τις πρακτικές και από εκεί και πέρα μπορεί να διαφέρουν και λίγο και τα μοντέλα εφαρμογής. Σε κάποια κράτη-μέλη, ακόμα και αν είναι πολύ συγκεκριμένη νομοθεσία και δεν είναι ε, δίκαιο ανταγωνισμού, ε, η αρχή ανταγωνισμού είναι αυτή η οποία το επιβάλλει και αυτές είναι οι πράσινες χώρες, η Ιταλία τουλάχιστον είναι μία εξ αυτών και μετά υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αρχές οι οποίες εφαρμόζουν αυτή την ομοθεσία. Αυτό είναι το ένα μοντέλο. Μετά, όπως σας είπα, μπορεί να υπάρχει κάποια προσαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού. Είχαμε μια πρόσφατη αλλαγή στη Φιλανδία, για παράδειγμα, ή δίκαιο ανταγωνισμού, το οποίο είναι ακόμα είναι ήδη ενισχύ και βασίζεται στην εξέταση της οικονομικής εξάρτησης μεταξύ των συμβαλωμένων μερών και της αγοραστικής δύναμης. Ε, και για παράδειγμα αυτό είναι η λύση που επέλεξε η Γερμανία και εφαρμόστηκε προσφάτως σε μία υπόθεση ε, στην οποία υπήρχε προσφυγή κατά ε, ενός από τους μεγάλους λιανοπολιτές στη Γερμανία. Ίσως υπάρχει κάποιο σημαντικό δίκαιο το οποίο ενδεχομένω θα μπορούσε να εφαρμοστεί, αλλά πρέπει κανεί να προσφύγει στα δικαστήρια και όπω καταλαβαίνετε υπάρχουν διάφοροι περιοριστικοί κανόνε. Στη μελέτη απεδείχθη επίση ότι υπάρχουν κάποιες αθέμητες πρακτικές χωρίς να μπορεί κανείς να προσφύγει. Όλα αυτά τα θέματα συζητώνται. Τι οδήγησε την Κομισιό στο να ενεργήσει έτσι και να δημοσιεύσει αυτή την ανακοίνωση. Πρώτα απ' όλα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει ο νόμος περί ανταγωνισμού με τρόπο αποτελεσματικό το άρθρο 1.1 και 1.2 τι συνθήκες αναφέρονται τέτοιου θέματα, αλλά ίσως η εθνική νομοθεσία κάθε χώρας να έχει ε, κάποιες ε, περαιτέρω ιδιαιτερότητες. Επίσης δεν υπάρχει εναρμονισμός στα πλαίσια του άρθρου και των 2. Και ίσως τα κράτη-μέλη να έχουν τέτοιου είδους διατάξεις και προβλέψει σε περίπτωση τέτοιου είδους αθέμητων πρακτικών, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Η πρωτοβουλία για την εφοδιαστική αλυσίδα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και το τονίζω και το ξανατονίζω και θα πρέπει το θέμα αυτό να το χειριστούμε με τρόπο ευέλικτο αλλά υπάρχουν και σε θέματα αυτά των αφέμητων πρακτικών κάποιες αδυναμίες, κάποια κενά που έχουν σχέση με την ε, εφαρμογή τους και αυτό είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους θέλουμε εμείς ε, να ολοκληρώσουμε την παρουσία της ανακοίνωσης αυτής και πιστεύουμε ότι καλό θα ήταν επίσης να τονίσουμε ότι όντως υπάρχει καλύτερη κατανόηση τώρα για τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με νομοθετικό μέσον. Αλλά στα πλαίσια της εναρμόνισης καλό θα είναι να πούμε ότι υπάρχει γενικότερη συνένεση για τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα των ειδών διατροφής. Τώρα όσον αφορά την εφαρμογή. Πιστεύω ότι η σωστή εφαρμογή είναι πάρα πολύ σημαντική σε εθνικό επίπεδο. Έγιναν συζητήσεις επίσης για το γιατί η Κομισιό δεν πρότεινε μία πιο εύρωστη ε, πρόταση, παρά μόνο μία ανακοίνωση, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, όπως, όπως αφήνισε προηγουμένως, το θέμα είναι θέμα εσωτερικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι κάποιες αθέμητες πρακτικές ε, εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο με διαφορετικές νομοθεσίες. Η τάση είναι να προσπαθήσουμε να διεργήσουμε κάτι το καλύτερο στα πλαίσια του νέου νομοθετικού πλαισίου. Όσον αφορά την εφαρμογή και νομίζω ότι δεν θα δεν ήταν εύκολο να βρούμε μια λύση που να ισχύει με τον ίδιο τρόπο για όλους. Νομίζω ότι με τους χάρτες που σας έδειξα καταλάβω ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μια ενιαία λύση. Τελικά και πάρα πολύ σημαντικό. Η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ νέα. Την επεξεργαζόμαστε εδώ και λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μας αποδείξει ότι είναι εποφελής, χρήσιμη και γι' αυτό προς το παρόν περιοριζόμαστε σε ανακοίνωση. Τώρα, τι κάνουμε στα πλαίσια αυτής της ανακοίνωσης. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι απευθυνόμαστε σε χώρες όλες σε θέματα εμπορικών πρακτικών. Βάση σε τρεις άξονες. Πρώτα απ' όλα έχουμε αυτή την πρωτοβουλία ε, την εφοδιαστική αλήθεια. Δεύτερον, τις βέλτιστες πρακτικές. Τρίτον, αποδοτική εφαρμογή οδηγία σε εθνικό επίπεδο. Διότι ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι θα υπάρχει μια κοινοτική αρχή εφαρμογής της πρωτοβολίας σε κάθε χάρα μέλος είναι αυτή που πρέπει να αξιολογήσει πώς εφαρμόζεται αυτή η πρωτοβουλία τη δική της επικράτεια. Κάτι που δεν ανέφερα σχέση με την πρωτοβουλία εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ότι σε κοινοτικό επίπεδο ενθαρρύνουμε στην ανακοίνωση μας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προσυπογράψουν να συμφωνήσουν. Μας απασχολεί το τι θα κάνουν και οι ΜΜΕ στην εφοδιαστική αλυσίδα, διότι τους αφορά πολύ το σύνολο των ε, θέμητων πρακτικών. Και αυτός είναι ένας από τους στόχους αυτών που πρότειναν αυτή την πρωτοβουλία. Ποιες είναι το με αυτό προδιαγραφές σε κοινοτικό επίπεδο. Προανέφερα, χωρίς να μπορέσω να μπω σε λεπτομέρειες, ότι έχουμε συνένεση και αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ζητήσαμε από τα κράτη-μέρη να εξετάσουν εάν το ρυθμιστικό τους πλαίσιο συνάδει με αυτές τις αρχές. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να δούνε ποια είναι η κείμενη νομοθεσία, όχι σε θέματα πεδιοφαρμογής, αλλά και κυρίως όσον αφορά το περιεχόμενο των πρακτικών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται, διότι όπως και σε πολλούς άλλους τομείς υπάρχει τάση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό να είναι πάρα πολύ επαχθείς οι κανόνες. Επίσης τονίζεται η... πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ένα αποτελεσματικό αποτρεπτικό σύστημα και είναι επίσης σημαντικό το σύστημα να μπορεί στην πράξη να δουλεύει σωστά. Να ισχύει εδώ η αρχή του απορρίτου, να μπορεί κανείς να είναι σε θέση να κάνει έρευνα σε περίπτωση προβλημάτων όταν εφαρμόζει τέτοιου είδου αθέμητε ε, πρακτικές. Υπάρχει και αυτό το οποίο ονομάζουμε συντελεστής ε, φόβου, εάν κανείς προστρέχει σε τέτοιου είδου πρακτικές. Και ξέρουμε πολλές φορές ότι όταν το πιο αδύναμο σκέλος μιας ε, σχέσης καταγγείλει μια τέτοια πρακτική, φοβάται ότι θα του επιβληθούν αντίπεινα. Προσπαθούμε αυτή την κατάσταση να διευθυντήσουμε και να μπορούμε να ερευνούμε σε περίπτωση τέτοιων προβλημάτων. Συμπερασματικά και συνοπτικά. Τι μάθαμε για τα έρχεται της μελέτη και τι συμβαίνει τώρα. Ένα χρόνο μετά την ε, εκτίμηση, ζητήσαμε να γίνει μια μελέτη σε σχέση με την πρωτοβουλία αυτή και το τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Θα αναλύσουμε περισσότερο το τι γίνεται με την εθνική νομοθεσία. Θα ζητήσουμε τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν βέλτιστες πρακτικές. Θα συντονίσουμε το τι ακριβώς γίνεται σε κάθε χώρα και χώρα και θα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη για να δούμε πώς αξιολογούν τα ίδια τα κράτη-μέλη, τα συστήματά τους και θα σας αναφέρουμε μετά τα τελικά συμπεράσματα αυτής της μελέτης και σας και στο Συμβούλιο. Το 2015 θα συντάξουμε και κάποιες συστάσεις για να δούμε εάν σε κάποιες περιπτώσεις συνιστάται περαιτέρω κοινοτική δράση. Ελπίζω ότι σας έδωσα να καταλάβετε το περιεχόμενο της μελέτης και της ανακοίνωσης της Επιτροπής και είμαι στη διάθεσή σας βεβαίως για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση θέσετε. Um, Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε και θέματα που αφορούν την Επιτροπή ίντε. Λοιπόν, επειδή πραγματικά ο χρόνος μας πιέζει, όποιος θέλει να κάνει ερώτηση από τους κοιόδης ή μπορεί να το κάνει, αλλά πάρα πολύ σύντομα. Έχουμε 7 λεπτά στη διάθεσή μας. Ξεκινάμε με τον κύριο Τζάκεβιτς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για περίπλοκα θέματα και πολύ δύσκολα θα τα καλύψουμε σε λίγα λεπτά. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Επιτροπής για αυτήν την παρουσίαση των βασικών πρακτικών του ανταγωνισμού του τομέα. Ξεκινάει η συζήτηση και πρόκειται για μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας με σκοπό να κάνουμε έναν απολογισμό κοινών σημείων και κοινά αποδεκτών προτάσεων έτσι ώστε να αποτρέψουμε τέτοιου είδους ε, πρακτικές του ανταγωνισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες πρακτικές του ανταγωνισμού οι οποίες πλήττουν τον τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να τις ε, περιορίσουμε έτσι ώστε να υπάρχει ενίσχυση του διασυνοριακού εμπορίου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερες επενδύσεις και πιο υγιής ανταγωνισμός. Για μένα είναι πολύ σημαντικό όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε αυτήν την διαδικασία. Εγώ θα εξετάσω πάρα πολύ προσεκτικά όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν. Έχουμε την έκθεση της κυρίας Μπίλτ, του κυρίου Ντεγιόγκ, Υπάρχουν ήδη δράσεις ε, οι οποίες ε, έχουν ξεκινήσει για τον ορισμό αυτών των αθέμητων πρακτικών, παραδείγματος χάρη και τον Ιανουάριο του 2012, η έκθεση για τον τομέα αυτό των τροφίμων αναφέρει ότι χρειάζεται ρυθμίσεις, έλεγχος και κυρώσεις. Το 2013 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πράσινη βίβλος για αυτές τις πρακτικές του ανταγωνισμού. Το 2010, όπως είπε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, υπήρχε το κείμενο για την διατροφική αλυσίδα, τις αδυναμίες και τα προβλήματα. Και επίσης μιλούσε το κείμενο αυτό για το θέμα της αυτορύθμισης ιδιαίτερα για το τομέα της λιανικής πώλησης. Όμως, πραγματικά ο δεσμευτικός χαρακτήρας αυτού του συστήματος ισχύει και εφαρμόζεται μόνο για αυτούς που έχουν υιοθετήσει το σύστημα. Σήμερα πρέπει σαφώς να δούμε ευρύτερα το θέμα και τις περιπτώσεις ε, βεβαίως B2B όχι μόνο δηλαδή το λιανικό εμπόριο. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, δεσμευτικές ή όχι. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύψουμε όλες αυτές τις πρακτικές. Παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα και πάρα πολλές προτάσεις, βλέπουμε ότι η προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική από τη μία χώρα στην άλλη και το θέμα γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχουν μηχανισμοί εφαρμογής των διατάξεων και των κειμένων που υπάρχουν για την πάταξη και τον περιορισμό των αθέμητων πρακτικών. Δεν υπάρχει εναρμόνιση. Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για τον τομέα της διατροφικής αλυσίδας. Είναι επίσης εδώ ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα προτάσεων της Επιτροπής. Διότι έχω την εντύπωση ότι αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί δεν αρκεί να ζητήσουμε από κάποιους προαιρετικά και αν το επιθυμούν να τηρήσουν κάποιες κάποια μέτρα και κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικά κείμενα, υποχρέωση τήρησης κάποιων προδιαγραφών και κυρώσεις. σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουν λοιπόν οι αθέμητες αυτές πρακτικές, θα πρέπει να τις περιορίσουμε, να υπάρξουν κυρώσεις και να σταματήσουν οι καταχρήσεις οι οποίες συνεχίζονται. Είναι πολύ σημαντική η αποστολή μας. Θα πρέπει να ξαναδούμε τις πολιτικές, τους τομείς, την εναρμόνιση της υπάρχουσας ε, νομοθεσίας και συνόλου ρυθμίσεων και συμπερασματικά θα ήθελα να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις η εκπρόσωπος της Επιτροπής. Η έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά το λιανικό εμπόριο του Δεκεμβρίου του 2013 έκανε μια έκκληση προς την Επιτροπή για την εξέταση των αναγκών και την εφαρμογή των κειμένων που υπάρχουν έτσι ώστε να περιοριστεί το πρόβλημα. Το αναφέρατε αυτό, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς κάνατε μέχρι σήμερα έτσι ώστε να μειωθεί η ανησυχία και η αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά. Δεύτερη ερώτηση που απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει δυνατότητα υιοθέτηση δράσεων αποτελεσματικών έτσι ώστε αυτή η μάστιγα των αθέμητων πρακτικών που πλήττουν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παταχθεί. Και νομίζω ότι εδώ εκπροσωπώ και πολλούς άλλους ε, Ευρωπαίους επιχειρηματίες. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την αγορά στην ενδεχόμενη αυτορύθμιση. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε προαιρετικά και αν το επιθυμούν οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν κάποιους κανόνες. Σκοπός μας είναι η πάταξη αυτού του φαινομένου αλλά και η αποτροπή του. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή ξεκινήσαμε καθυστερημένα, μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Λοιπόν, ή θα επανέλθουμε αύριο το πρωί στο τέλος της ημερήσιας διάταξης στο θέμα αυτό. Θα ξαναδώσω το λόγο στους σκιώδες και θα δω αν χρειάζεται όμως αύριο στο τέλος της ημερήσιας διάταξης να επανέλθουμε θα το κάνουμε. Εγώ θέλω πραγματικά σε πέντε λεπτά να δώσω το λόγο στους συντονιστές που θα συνεδριάσουν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ που δεν θα μπορέσει να έρθει σήμερα και μου ζήτησε να παρουσιάσω τις παρατηρήσεις της. Χαίρεται που ε, η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων βρίσκεται στις προτεραιότητές μας και θα ήθελε να ζητήσει από τον κύριο Γιάβκοβιτς ε, να συνεχίσει να εργάζεται επί του θέματος και να συνεχίσει τα καλά αποτελέσματα ε, συμπεριλαμβανομένων και των όσων έχει να προσθέσει η ίδια η κυρία Κοράτσα Μπίλτ για μια πιο αποτελεσματική και δίκαιη αγορά λιανικών πωλήσεων ή το πρόγραμμα δράσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την λιανική αγορά και το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το B2B, το business to business. Ε, υποστηρίζει την πρωτοβουλία για την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, καθώς επίσης και τονίζει ότι θα πρέπει να ε, έχουμε θεμητές εμπορικές πρακτικές, τις σχέσεις ε, μεταξύ επιχειρήσεων. Είναι κάτι το οποίο ε, προχωρήσαμε τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος. Αρχικώς υπήρξε άρνηση και τώρα έχουμε αρχίσει να προχωρούμε σιγά σιγά και πιστεύει ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα σε συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. και θα πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε με έναν επικοδομητικό διάλογο όπως αυτόν που έχουμε με τους ενδιαφερομένους. Ενθαρρύνει επίσης όλους τους ενδιαφερομένους να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αλλά και στη δημιουργία αντίστοιχων αντίστοιχης πλατφόρμας σε εθνικό επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ε, να επιδείξουν υπευθυνότητα και να κάνουν τα πάντα με διαφάνεια. Υπάρχει επίσης η ετήσια στρογγυλή τράπεζα λιανικών πολίσεων, την οποία έχει συστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ένα φόρουμ που θα συζητά και θα αξιολογεί την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Η κυρία κορατσα Μπίλτ προσβλέπει στην επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή και με τους υπόλοιπους και οδησηγητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μας μένει πολύς χρόνος. Τέσσερις ερωτήσεις θέλω να κάνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και για την παρουσίασή της και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, διότι αναφέρθηκε σε πολλά από τα στοιχεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ κι εγώ. Ε, πρέπει να πω ότι είμαι μάλλον επιφυλακτική ε, για αυτό το εθελοντικό σύστημα. Είναι μεν μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, αλλά στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγεται ότι στην πρωτοβουλία δεν συμμετέχουν οι γεωργοί, δεν συμμετέχουν οι εκπρόσωποι του ε, τομέα του κρέατος. Τι ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμμετέχουν τότε. Πόσοι μικροί ενδιαφερόμενοι ε, συμμετέχουν σε αυτή την ε, εθελοντική πρωτοβουλία από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Μία ακόμα ερώτηση. Ευρωπαϊκή Ένωση. το το θέμα τα περιθώρια ευελιξία. Έχω ξαναθέσει αυτή την ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν μου απάντησε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει στατιστικά στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε τι ε, περιθώριο έχουν ε, τα κράτη-μέλη. Και εδώ έρχομαι στην τρίτη ερώτησή μου. θα θέλαμε μια πιο λεπτομερή ανάλυση για τις συνέπειες των αθέμητων εμπορικών πρακτικών για τον τελικό καταναλωτή. Και ένα τελευταίο σχόλιο. που έχει σχέση με ισότιμη αντιμετώπιση στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν και εθνικοί φορείς και παραγωγή, αλλά και άλλοι. και μπορούν να εφαρμοστούν διάφοροι κανόνες. Ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πώς έχει κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο Ρόμπερτ. Ευχαριστώ, Βίκη, πολύ σύντομα. Είμαστε εδώ ενώπιον ενό προβλήματο που δεν νομίζω ότι θα επιληθεί. Υπάρχει ουσιαστικά ανισότητα μεταξύ των μερών που εμπλέκονται, δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις όμιλοι από τη μία και από την άλλη μικρές επιχειρήσεις ή φορείς. Στη Γαλλία προσπαθούμε να βρούμε λύση, αλλά πολύ φοβάμαι ότι η λύση δεν θα βρεθεί εύκολα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πρώτον, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ανισότητα και τα διαφορετικά μεγέθη, όντως υπάρχει το πρόβλημα του φόβου, δηλαδή αυτό που αποτρέπει τις μικρές επιχειρήσεις να στραφούν κατά μιας μεγάλης, ενός μεγάλου ομίλου. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Όλα αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ και χρόνια Δηλαδή να βρούμε εναλλακτικού τρόπους για την εξέβρεση λύσεων, εκτός δηλαδή δικαστικού συστήματος. Φοβούνται οι μικρές επιχειρήσεις να προσφύγουν στα δικαστήρια. Με διαμεσολαβητές παραδείγματο χάρη. Ενδεχομένως αυτό δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βρεθούν λύσεις και να βρεθεί κάποιος διακανονισμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Ερωτώ και την Επιτροπή και τον εισηγητή. Αυτού του είδους δηλαδή η διαμεσολάβηση μήπως θα μπορούσε να αποτελέσει λύση. Τώρα, οι 28 εμπειρογνώμονες έκαναν κάποιες συστάσεις, μία εξ αυτών είναι ενδιαφέρουσα κατά την άποψή μου, γιατί να μην προετοιμάσουμε ένα κατάλογο των λεγόμενων μαύρων ή γκρίζων, των αθέμητων πρακτικών δηλαδή. Σήμερα δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε ένα νομοθετικό μέσο εργαλείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά τουλάχιστον αφού υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε αυτό το κατάλογο αθέμητων πρακτικών, τον λεγόμενο μαύρο ή γκρίζο κατάλογο, να παρατηρήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και να τα καταγράψουμε. Ίσως αυτός θα μας βοηθούσε λίγο ε, στην αποτελεσματική μας δράση. Ο κύριο Τάντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο και νομίζω ότι άπτεται ενό ε, πολύ σημαντικού θέματο για να εγγυηθούμε προστασία των καταναλωτών και σωστή σχέση μεταξύ του εφοδιασμού των τροφίμων και των παραγωγών τροφίμων. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, κυρίω στον γεωργικό κόσμο και κυρίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Μιλά πολύ γρήγορα. Α, συγγνώμη, απλώ δεν έβγαινε η διερμηνία. Α, συγγνώμη. Ε, είναι πάντα αυτό. Πρέπει να μιλάμε αργά, αλλά πρέπει να τα λέμε και στα γρήγορα. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να μιλάω αργά, αλλά να τα πω σύντομα. Θα πω λιγότερα. Έλεγα λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι αφενός ε, διαπιστώνουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση των, μικρών, ε, των μεγάλων συγγνώμη, επιχειρήσεων διανομής, ε, αρκεί να δει κανείς ε, ε, σε οποιαδήποτε πόλη της Ευρώπης ότι έχουμε τις ίδιες εταιρείε που διανέμουν τα προϊόντα σε όλη την Ευρώπη, είτε στην Ιταλία, είτε στη Γαλλία, είτε στη Γερμανία, λίγο πολύ οι ίδιοι ισχυροί είναι, οι οποίοι όπως έλεγε και ο συνάδελφος ε, Ροσφόρ ε, ε, πριν, έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπορική ισχύ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό, ώστε στο μέλλον η αποτελεσματικότητα της εμπορικής διανομής να μην είναι ευθύνη των παραγωγών, διότι πολλές φορές η αποτελεσματικότητα της, διαμονε... Ε, διανομής ήταν εις βάρος των παραγωγών και απλώς οδηγούσε σε μείωση της τιμής. Και έχω την ε, εξή ερώτηση να θέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από αυτές τις ε, πρακτικές που θεωρούνται αθέμητες υπάρχει και η δυνατότητα των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν το εμπορικό του σήμα για να διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα ε, που έχουν ζητήσει από άλλες εταιρείες παραγωγής. Αυτό φυσικά επηρεάζει πάρα πολύ τις επιλογές της αγοράς, δεν εγγυάται τίποτα στον καταναλωτή και κυρίως στερεί από τους παραγωγούς ε, το ε, στοιχείο της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων τους. Θα ήθελα να ξέρω εάν αυτό είναι μία από τις πρακτικές που θα ήθελε να αναλύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να προβλέψουμε να γίνει κάτι περαιτέρω στο θέμα αυτό και να μην έχουμε απλώ μια εθελοντική πρωτοβουλία σαν αυτή που μας παρουσιάστηκε. Ευχαριστώ. Μπορούμε πάντα, επανέλθουμε το όντως, και εγώ διαπιστώνω ότι είναι αργά, είναι 6 ευχαριστώ για το σχόλιά σας. Πάρα πολύ σύντομη, δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες. Κάποιο πρόβλημα έχει η διερμηνία, λέει η Πρόεδρος. Δεν ακούγεται. The channels Okay, now we're hearing the English. Thank you. Thank you. Λέγα, um, Έλεγα, λέει η πρόσωπος της Κομισιόν ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε, με λεπτομέρειες. Μπορείτε να επανέλθετε αύριο το πρωί για να μας απαντήσετε λεπτομερώς ερωτήσεις. Το δέχονται αυτό οι, οι συνάδελφοι καθώς και ο συγγετής. διότι έχουμε τουλάχιστον μισή ώρα ερωτήσεις εκ μέρους των μελών και θα ήθελε σε κάποιες από αυτές να απαντήσει η Κομισιό. Αύριο στις 11 παρα 10, στις 11 και 10 μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ή θέλετε γραπτές απαντήσεις, ο εισηγητής αποφασίζει αύριο. Tomorrow is good. Έχει καλός. Αύριο λοιπόν. Ε, κύριε Ροσφόρ, θα είστε εδώ αύριο? Εδώ θα είμαι, αλλά την ίδια στιγμή θα έχω κάποια άλλη συνεδρίαση. Ε, η Κομισιόν μπορεί. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά, πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και την ευελιξία σας. Και τώρα περνούμε στην συνεδρία των συντονιστών. Thank